Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την αφήξω τον πρέσβη για την παρουσία του εδώ. Και βέβαια, εμείς θα πάμε στον Πενοσάιρες και θα συμμετάσχουμε σε αυτό το κοινοβουλευτικό φόρουμ της ομάδας των 20. Το περιμένουμε πώς και πώς. Προχωράμε γιατί είμαστε υπό μεγάλη πίεση χρόνου. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε ευθύ αμέσω στο σημείο 11 τη μερσιά διάταξη, που είναι ανταλλαγή απόψεων για τι εμπορικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία τη Νοτιοαφρική. Να καλωσορίσω ε, τους εκπροσώπους, ε, του, τα μέλη της με την προσωπία λοιπόν από την πρεσβεία της ε, Νοτιοαφρικής Ο πρέσβης νομίζω, ο ίδιος... Ε, Again, I apologize. Βάσος Σανκού είναι εδώ. If not, then uh, you can correct me later. Ελπίζω να το πρόφερα σωστά, αλλιώς διορθώστε με. Επιταμελής αντιπροσωπεία της ΙΝΤΑ θα μεταβεί στην Νότια Αφρική στα τέλη Οκτωβρίου για να δει πώς προχωρά η υλοποίηση της ε, οικονομικής εταιρική σχέσης. Δύο χρόνια πάνε από τότε που τέθηκε σε ισχύ. Θα συζητήσουμε επίσης ε, με τους ομολόγους μας και τα ε, μερή ζητήματα. και τις εμπορικές μας σχέσεις. Πέρασε καιρό που είχαμε συζήτηση για τα θέματα των εμπορικών αυτών σχέσεων στην Επιτροπή μας. Ε, δεν θα καθυστερήσω, αλλά θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρια Σκόλα, που είναι η αναπληρώτρια τμήματάρχη, μάλλον επικεφαλής μονάδας για τις οικονομικές εταιρικέ σχέσεις. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτήν την δυνατότητα να μιλήσω ενώπιόν σας τη στιγμή που ε, ε, διανύουν η σχέση ε, με την, Νότια Αφρική μια ιδιαίτερα μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις. Η Νότια Αφρική είναι στρατηγικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός τη Αφρικής, αλλά η οικονομική και κοινωνική διάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος επενδυτής με 78, στην ε, Νότια Αφρική ε, με 78% ε, όσον αφορά τις και 30% όσον αφορά τις εμπορικές ροές. Μετά έρχονται η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε με 18 και 7% αντίστοιχα. Η Νότια Αφρική βεβαίως συμμετέχει στην ΣΑΝΤΕΚ ΕΙΠΑ μαζί με την Αμίμπια, τη Μοζαμβίκη, την Ποτσουάνα και τη Σουαζιλάνδη που εφαρμόζεται εδώ και δύο χρόνια πλέον. Η Νότια Αφρική βεβαίως αποτελεί μια ιδιαίτερη διάζουσα περίπτωση σε αυτή την ΕΙΠΑ, γιατί αντίθετα από, τις, τα άλλα μέλη ΣΑΝΤΕΚ δεν έχει πλήρη πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το άνοιγμα της αγοράς είναι περίπου στο 94% γενικά, ενώ η, ε, το, ε, η αγορά της Νότιας Αφρικής έχει ανοίξει ε, περίπου γύρω στο 84% για προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια σημεία τριβής, κυρίως όσον αφορά τα πουλερικά εξαγωγές πουλερικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Νότια Αφρική. Δεν είναι πρώτη φορά που συζητιέται το θέμα αυτό στην Επιτροπή σας, αλλά θα ήθελα να κάνω μια μικρή ε, σύνοψη. Το 2015 ε, η ε, ε, Νότια Αφρική επέβαλε ειδικού φόρους anti-dumping για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία ισχύουν ακόμα και δεν διαφορούμε τα μέτρα αυτά. Το 2016 όμως η Ευρωπαϊκή, η Νότια Αφρική λόγω της γρήπης των πτηνών κατήργησε τις ε, εισαγωγές ε, από 8 ε, χώρες, από τις οποίες μονάχα για την Ισπανία έχουν αρθεί οι απαγορεύσεις, ενώ εδώ και ένα χρόνο δεν υπάρχουν πλέον κρούσματα αυτής της ασθένειας. Τον Σεπτέμβριο του 2018, φέτος δηλαδή, η Τελωνιακή Ένωση της Νότιας Αφρικής Σακού επέβαλε ε, ρήτρα ασφάλειας 35,3% ε, για τα ευρωπαϊκά πουλερικά. Βεβαίω υπάρχει μία ε, διάταξη στα πλαίσια του ΣΑΝΤΕΚ που προβλέπει ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, αλλά εμείς θεωρούμε ότι δεν, έχουν, δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο το μέτρο αυτό και ε, θεωρούμε ότι ε, σύμφωνα με τους, ε, τις διατάξεις η διατάραξη της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να απορρέει από την ΕΠΑ απευθείας και εδώ δεν είναι αυτή η περίπτωση. Ε, επίσης, ε, λόγω και των λοιπών μέτρων έχουν ε, υποχωρήσει κατά πολύ και οι, γενικότερα οι εξαγωγές προς την Νότια Αφρική, πράγμα ε, πράγμα που σημαίνει ε, ότι ε, η θέση, το κενό που άφησαν οι εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλύφθηκαν από γηγενείς παραγωγούς, αλλά από τη Βραζιλία και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Επίσης, προσπαθούμε να βρούμε επικοδομητική λύση με τους ε, ε, ομολόγους μας της ε, Νοτιού Αφρικής. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει αποστολή υψηλού επίπεδου στη Νότια Αφρική για να συζητηθεί το θέμα αυτό σε μια προσπάθεια επίτευξης ε, συμβιβασμού. Στις 15 Νοεμβρίου επίση, θα λάβει η χώρα εδώ στις Βρυξέλλες διάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και νότια Αφρικής και βεβαίω ευελπιστούμε ότι θα έχουμε προχωρήσει αρκετά στην επίλυση των θεμάτων αυτών πριν τη διάσκεψη κορυφή. Επίσης η Επιτροπή Εμπορίου και Ανάπτυξης ε, που είναι υψηλού επίπεδου για την επιτήρηση της ΕΕ θα συνεδριάσει με το ίδιο θέμα τον Φεβρουάριο του 2019 θα έχουμε ε, την ε, το πρώτο συμβούλιο σε επίπεδο υπουργών στο Cape Town Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΠΑ ΣΑΝΤΕΚ. Επίσης, ευελπιστούμε ότι όταν θα πάει στη Νότια Αφρική ε, η αποστολή της Επιτροπής σας θα βοηθήσει στην άβλυνση των προβλημάτων ε, θα υπάρξει βεβαίως και τεχνική ενημέρωση πριν φύγετε στις 24 Οκτωβρίου και αν θέλετε τότε θα σας δώσουμε οπωσδήποτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Ευελπιστώ ότι την επόμενη φορά που θα σας μιλήσω θα είμαι ελπίζω σε θέση να σας δώσω και πιο θετικά νέα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τον μόνιμο ε, εισηγητή, την μόνιμη, Νάντια Χέρσο, για το θέμα, Η εισηγήτρια μόνιμη της ΙΝΤΑ. Αξιότιμε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εισαγωγικέ της παρατηρήσεις που ήταν μια επισκόπης κατάστασης. Ε, η οικονομική εταιρική σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική και για τις εμπορικές προτιμήσεις ε, που ε, έχουμε αποφασίσει να συνεχίσουμε μετά την Κοτονού με τις χώρες και έχουμε και με πολλές άλλες χώρες. Υπάρχουν πάντως ασημέτριες και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα γενικό πρότυπο για την ε, εποχή μετά το Κοτονού και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτή η ε, συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί και η εφαρμογή να βελτιωθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει πρόοδος στην Νότια Αφρική και στην ευρύτερη περιοχή βέβαια. Βλέπουμε δείγματα πρόοδου σε αρκετούς τομείς σε ό,τι αφορά παραδείγματο χάρη την ενοποίηση τη κυκλοφορία, ε, ε, το West Africa Cable System, επίση ένα σημαντικό ε, βήμα προόδου για να υπάρχει γρήγορο ίντερνετ στην όλη περιοχή και το roaming επίση είναι ένα project το οποίο προβλέπεται στην ευρύτερη περιοχή και θα βοηθήσει όχι μόνο την κοινωνία αλλά και την οικονομική πρόοδο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις σχέσεις ε, με την ε, Νότια Αφρική και την περιοχή, υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, το είπατε κι εσείς ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πράγματι δεν είναι απλή η περίπτωση με την κρυπτών αλλά μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή έχει να κάνει και με την έλλειψη των, της συμμετοχής από τους φορείς και των πολιτών. Αυτό είναι εμφανές. Υπάρχει αυτή η έλλειψη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ακούσω την Κομισιόν ε, τι κάνει στις συνομιλίες της και πώς φροντίζει να σημειωθεί πρόοδος και σε αυτό το πολύ κομβικό σημείο για να έχουμε μεγαλύτερη πρόοδο. Και επίσης ε, η ε, στενή σύνθεσμοι με την τοπική οικονομία, κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Θα με ενδιαφέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσω αν στον τομέα αυτό έχουν σημειωθεί θετικές εξελίξεις ε, και φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε και στην επίσκεψή μας εκεί στα τέλη Οκτωβρίου ή το αργότερο εδώ που θα έχουμε τη διάσκεψη κορυφής της Βρυξέλλες σίγουρα μπορούμε να ενημερωθούμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Έχουμε τους σκιώδης τώρα. Θα πάρουν το λόγο. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Αν είναι εδώ θα πάρει το λόγο ο κύριος Γκαμπριέλ Μάτο εκ μέρους της ομάδας του ΕΛΚ. Δεν τον βλέπω τον κύριο Μάτο. Σε ποιον να πάω? Να πάω στους ελιστές και δημοκράτες και στον κύριο Γιώχιμ Σούστερ. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με την ε, ε, άποψη της εισηγητρίας ότι είναι σημαντική αυτή η συμφωνία και επομένως μας ενδιαφέρει να είναι και επιτυχής η εφαρμογή. Βέβαια υπάρχουν και κάποια επίμαχα σημεία τη συμφωνία. Δεν είναι εμπορική μόνο η συμφωνία αυτή. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ στρέφομαι στην Κομισιόν για να ακούσω τι γίνεται με τα άλλα σκέλη, την εφαρμογή των άλλων σκελών τη συμφωνία, ό,τι αφορά ε, την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και εμπορικής σχέση. Ε, σχέση. Ε, γιατί θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία, θέλουμε να ε, τηρηθούν οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη ε, κτλ. Εκεί Πώς πάει η εφαρμογή. Και αυτή είναι μια ε, σημαντική ερώτηση που και εγώ θα ήθελα να αναφέρω, πως και η συγγητρία. Τι γίνεται με τη συμμετοχή των οργανώσεων και των πολιτών. Νομίζω ότι υπήρχαν κάποιες θετικές εξελίξεις, προχωρά αυτό, βελτιώνεται η κατάσταση, υπάρχουν δυσκολίες θα ήθελα να πείτε πώς έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και επειδή μιλήσατε και για ε, το Υπουργικό Συμβούλιο ΣΑΝΤΕΚ ε, και Ευρωπαϊκή Ένωση το Φεβρουάριο, τι γίνεται με την, προπαρασκευή, την πρώτη ε, προπαρασκευή υπήρξε ένα θέμα, εντάξει δεν μπορούμε να το δούμε, ε, δεν μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες ακόμη, αλλά αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια πράγματα, κάποιες προφορίες για το θέμα. Ο κύριος David Campbell Bannerman, ECR δεν είναι εδώ, άρα θα ακούσουμε τον κύριο Σόλτς από την ΚΟΕ. Ούτε αυτός είναι εδώ. Η κυρία Χάουταλα μήπως είναι εδώ, ω πρασίνους. Ούτε και αυτή είναι εδώ. E Υπάρχει κάποιος άλλος που θα θέλει να το λόγο, παρακαλώ. Κανείς. Δεν βλέπω λοιπόν άλλου συναδέλφου. Πριν να δώσω και πάλι το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διευθύνση Εμπορίου, θα ήθελα να ζητήσω από το... την αυτή εξοχότητα τον πρέσβη τη Νοτιού Αφρική, τον κύριο Μπάσο Σανκού, να μα παρουσιάσει τη θέση του κράτου του. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμούμε ιδιαίτερα στην ευκαιρία που μας δίνετε να σας έχουμε αυτή τη συζήτηση, διαζώσεις για τη συνεργασία της Νοτιάς Αφρικής με την, με τις, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σημαντικό εμπορικό εταίρο για πολλά χρόνια για την Νότια Αφρική και επιθυμούμε αυτό να συνεχίσει. Ιδιαίτερα τώρα, που έχουμε εμβάθυνση της δημοκρατίας στη Νότια Αφρική και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις στην οικονομία. Τώρα ακριβώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εταιρική μας σχέση και η αμοιβαία συνεργασία. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Νότια Αφρική πιστεύει βαθύτατα στην πολυμερή διπλωματία πιστεύει ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ενωπής, ε, καλύτερης συνεργασίας, ε, ε, όχι μόνο γενικότερα της, της Νότιας Αφρικής, αλλά και γενικότερα της Αφρικής. Θεωρούμε πολύ σημαντική τη Συμφωνία Εμπορικής, ε, Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΣΑΝΤΕΚ. Δεν έχουμε ίσως ακριβώς την ίδια αντίληψη για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Πιστεύω ότι όλοι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτή την εμπορική συμφωνία όσο καλύτερα γίνεται στο πλαίσιο των κανόνων που έχουμε διαπραγματευτεί, του πλαισίου που αυτοί θέτουν. Όποιες προκλήσεις και να αντιμετωπίζουμε, αυτές πρέπει να τις επιλύουμε στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων. Έγινε αναφορά στο ζήτημα των πουλερικών. Πιστεύουμε ότι η Νότια Αφρική και η Σαντέκ ορθώς έχει ε, καθορίσει, εφαρμόσει αυτά τα μέτρα στο πλαίσιο των κανόνων του ΣΑΝΤΕΚ. Ήταν μια απόφαση των κρατών της ΣΑΝΤΕΚ Τα μέτρα αυτά υιοθετήθηκαν μετά από την πλήρη και ορθή διαδικασία που ακολουθήθηκε και στην οποία συμμετείχε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργεί κάποιες δυσκολίες και ότι είναι μια πρόκληση του γεγονός ότι έχουμε μια διάσταση απόψεων μεταξύ Νότιας Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα. Όπως ήδη ελέγχθη, συνεργαζόμαστε στενά για να λυθεί το πρόβλημα σε καμία περίπτωση αυτό δεν γίνεται με αρνητική πρόθεση από την πλευρά μας. Ε, ο Υπουργό μα έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώ προσπαθώντα να βρει λύσει, επιλογέ διαφορετικέ για να λυθούν συνολικά όλα τα προβλήματα και να προχωρήσουμε παραπέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, έχει εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να εφαρμοστούν διατάξεις της EPA. Και πράγματι υπάρχει αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από Γενική Διευθύνση Εμπορίου που συζητά τα ζητήματα αυτά στο Cape Town και ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουμε. Θα βρούμε. Έχουμε επίσης λάβει τις παρατηρήσεις των έξι κρατών που, για τις οποίες συνεχίζουν να υφίστανται τα μέτρα για την γρήπη των πουλερικών και έχουμε οργανώσει μια διάσκεψη στην Πρετόρια αυτή την εβδομάδα που επανεξετάζει το θέμα, την κατάσταση με αυτές τις έξι χώρες. Θεωρούμε πολύ σημαντική την επιτυχία αυτής της οικονομικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης όχι μόνο γιατί είναι σημαντική αυτή αλλά επίση και γιατί δείχνει το δρόμο για τι μελλοντικέ μα οικονομικέ σχέσει. και μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρικής, Νότιας Αφρική, αλλά και γενικότερα με την Αφρική, με την Ήπειρο τη Αφρική. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και άλλα θέματα επιτάπητος, όπως για παράδειγμα το ζήτημα του Χάλιβα. Εδώ πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε μονομερός απόφαση έναντι της Νότιας Αφρικής. Όταν ζητήσαμε εξηγήσει, ακούσαμε την απάντηση ότι ήταν λάθος και ότι προσπαθεί να επιληθεί, όμως θα θέλαμε, θα θέλαμε να μην επαναληφθεί αυτή η ατυχής, αυτό το ατυχές παριστατικό στις σχέσεις μας στο μέλλον. Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και θα ήθελα να ενθαρρύνω τα μέλη της Επιτροπής σας να επισκεφθείτε τη Νότια Αφρική έτσι ώστε να έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση, έναν ευρύτερο διάλογο με τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών στη Νότια Αφρική και να βρούμε κοινέ λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι επιτέλους μετά από πέντε χρόνια θα μπορέσουμε να διοργανώσουμε σύνοδο κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νότιας Αφρικής στις 13 Νοεμβρίου τρέχοντος. Είμαι σίγουρο ότι και πριν ή και κατά τη διάρκεια τη Συνόδου Κορυφή θα βρεθεί ένα τρόπο να επιληθούν τα ζητήματα. Εάν δεν βρεθούν λύσει πριν τη Σύνοδο Κορυφή, είμαι σίγουρο ότι οι ηγέτε μα στη Σύνοδο Κορυφή θα έχουν μια δυνατότητα να τα συζητήσουν και να τα επιλύσουν. Ε, ε, νομίζω και απαντώντα και σε ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έθεσαν το ζήτημα, πιστεύω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τη συζήτηση αυτή ω μόνο μια εμπορική συνεργασία, αλλά και ω μια ευρύτερη πολιτική συνεργασία μεταξύ των σε Ένωσης και, των, για της χώρας μου που θα πρέπει να ε, εμβαθυνθεί και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια ισότιμη συνεργασία αυτών των δύο μερών. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ξαναδώσω τον λόγο στην κυρία Σκόλα VVG Trade. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, να ρωτήσω πρώτα μήπως υπάρχουν ερωτήσεις ε, από πλευράς των βουλευτών μας, ε, ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που καθυστέρησα λίγο, αλλά έπρεπε να είμαι και σε μια άλλη συνεδρία ταυτόχρονα. Εν πάση περιπτώσει δεν άκουσα από την αρχή τη συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι αυτό που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κατανοήσουμε είναι... Ε, θα ήταν ποια μπορεί να είναι η επίκτωση του Brexit ε, στις ε, σχέσεις μας. Έχετε κάποιες, ε, ε, κάποια ε, άποψη ή κάποια στοιχεία όσον αφορά την επίπτωση που μπορεί να έχει ο, το Brexit και στα ναυτιλιακά και στην βιομηχανία, στον τεχνολογικό τομέα. Ίσως και η Κομισιόν θα μπορούσε να απαντήσει ή να σχολιάσει το ίδιο θέμα. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ε, άμεση ερώτηση στην εξοχότητά σας, αν θέλετε να απαντήσετε και μετά βεβαίω ε, αν δεν θέλει, θα επανέλθουμε και στην DigiTrade. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όπως φαντάζεστε, παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία του Brexit. Παρατηρούμε ωστόσο ότι πρόκειται στην ουσία για ε, εσωτερικές διεργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπα και προηγουμένως εμείς έχουμε ε, ιδιαίτερες ισχυρές σχέσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αλλά και με πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακολουθούμε τις διαδικασίες και τις διαπραγματεύσεις στενά αναμένοντας να δούμε που θα καταλήξουν έτσι ώστε ε, να δούμε και ποιον αντίκτυπο θα έχουν και σε εμά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είναι γεγονός ότι δυνητικά μπορεί να προκύψουν ε, επιπλοκές ε, σε σχέση με τη δικιά μας χώρα. Παρακολουθούμε στενά πάντως. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Μακουλάδα. Perdón, empiezo. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε ε, εκπρόσωποι της ε, Νότιας Αφρικής. Εγώ είχα την ευκαιρία να πάω ε, στην χώρα σας πριν έρθω εδώ ως βουλευτής και πραγματικά είναι αδύνατο να επισκεφθεί κανείς την Νότια Αφρική και να μην την ερωτευτεί. Και εγώ την ερωτεύτηκα τη χώρα αυτή. Θα ήθελα να υψώσω τη φωνή μου εξ ονόματος πολλών όμως γεωργικών, παραγωγών γεωργικών προϊόντων που προβληματίζονται λόγω των φυτοϊγειονομικών ελέγχων ε, σε σχέση ε, με τις επεξεργασίες διαφόρων ε, προϊόντων όπως ας πούμε των σπεριδοειδών. Ξέρετε ότι μέσω της νέας συμφωνίας γίνεται δυνατή η εισαγωγή εσπεριδοειδών τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη που όμως ε, είναι ακριβώς και η περίοδος ε, ε, συγκομιδής και εμπορίας των μεσογειακών εσπεριδοειδών. Πρέπει να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και χαίρομαι που είναι εδώ η Κομισιόν και με ακούει, γιατί δεν ε, βλέπουμε, δεν έχουμε στοιχεία για την εξέλιξη των ε, εισαγωγών από την, ε, συγγνώμη, από την Νότια Αφρική για το 17 και το 18. Είναι γεγονός πάντως ότι πιέζονται οι Ευρωπαίοι παραγωγοί. Και επίσης είναι γεγονός ότι ειδικά για τα, ε, ε, για τα πορτοκάλια. Ε, από τη δική μας πλευρά υπάρχουν κάποιες ασθένειες τις οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν λόγω της απαγόρευσης χρήσης κάποιων φαρμάκων. Γι' αυτό λοιπόν στρέφομαι προς την Κομισιόν και ρωτώ πότε θα μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις καταστάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο. Ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Όχι, οπότε ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση των ερωτήσεων. Θα δώσω ξανά το λόγο στον κύριο Πρέσβη, αν θέλει να απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα και μετά θα δώσω το λόγο στη DigiTrade. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ που θίξατε, αγαπητή ε, κυρία, το θέμα των εσπεριδοειδών. Εδώ και πολλά χρόνια ε, ε, η Νότια Αφρική εξάγει εσπεριδοειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι γεγονός ότι εμείς έχουμε διαφορετικό ε, ημερολόγιο παραγωγής και εμπορίας. Μπήκαμε, μπαίνουμε στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν έχουν ήδη όταν έχει ήδη ξεκινήσει η εμπορία των σχετικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά από πλευρά των Ευρωπαίων παραγωγών. Όσον αφορά ε, τους φυτοϊγειονομικούς κανόνες, η Νότια Αφρική ε, προσπαθεί να συμμορφώνεται με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό της κοστίζει πάρα πολύ, κυρίως όσον αφορά την εξαγωγή εσπεριδοειδών, καθότι η έννοια ε, του, κινδύνου ε, για, του, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αυτού του καρπού είναι τελείως, οι διαπόψεις λέω είναι τελείως διαφορετικές. Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια λύση. Και δεν έχουμε πρόβλημα να επισκεφθούμε την IPPC που είναι εμπειρογνώμονες για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα επίσης να πω ότι βεβαίως είχαμε μια καλή χρονιά και μια καλή συγκομιδή στην Νότια Αφρική. Αυτή τη στιγμή έχουμε παρακράτηση μονάχα ενός CBS ε, και σε σχέση με άλλους εξαγωγούς ε, δεν ε, νομίζω ότι εμείς αποτελούμε σημαντικό κίνδυνο για την ενωσιακή αγορά. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Άσκολα για ε, εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, πολύ σύντομα, να απαντήσω σε ένα σχόλιο για την μετά το κοτονού κατάσταση και την ασυμμετρία. Ε, αυτή η αρχή αναφέρεται επαρκώς ε, σε όλες τις εμπορικές ε, ε, συμφωνίες. Η κατάσταση μετά το Κοτονού ή μάλλον στην ε, μετά το Κοτονού περίοδο δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτό το θέμα μετά την εκπνοή της Συμφωνίας Κοτονού ε, ε, θα υπάρξουν βεβαίως κάποιες ε, τεχνικές τροποποιήσεις. Ωστόσο, οι κύριες αρχές που αφορούν την ασυμμετρία δεν θα τροποποιηθούν όσον αφορά την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα έχει μια συνάντηση στην Ναμίμπια την 8η Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, όπου αναμένουμε ότι θα υπάρξει και ε, ε, συζήτηση για το θέμα και επίσης μια αντίστοιχη ε, συνάντηση ΣΑΝΤΕΚ σε υπουργικό επίπεδο. Το δουλεύουμε αυτό. Επίσης θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν κοινό μηχανισμό επιτήρησης που θα ε, ε, ασκεί επιτήρηση όχι μόνο για θέματα σχέσης ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία των σχέσεων μηδεν, μηδεν, μιας, μηδενός εξαιρουμένου, ούτε της βιώσιμης ανάπτυξης κλπ. Επίσης, έχουμε προγράμματα διάφορα 6 εκατομμύρια ευρώ για κάθε, έχουν δοθεί για κάθε ε, χώρα χώρα και για την υλοποίηση της συμφωνίας. Ε, προς ώρας ε, ακόμα συστήνουμε κάποιους ε, οργανισμούς ή θεσμούς που θα βοηθήσουν στην πλήρη υλοποίηση της συμφωνίας στο σύνολό της όσον αφορά το θεματολόγιο της κοινής, του κοινού Υπουργικού Συμβουλίου. Θα δώσω το λόγο ε, στον συνάδελφο Γιάνν Βίλεμ Φερχάιντεν που προετοιμάζει αυτήν την συνάντηση. Σας ευχαριστώ. Στις 9 Φεβρουαρίου θα γίνει αυτή η Υπουργική στο Cape Town και βεβαίως θα προηγηθεί μια προπαρασκευαστική συνάντηση της ε, ομάδας εμπορίου και ανάπτυξης που προβλέπεται στην EPA. Αυτό θα γίνεται την επόμενο μήνα στο Johannesburg. Δεν μπορώ να προκαταλάβω βέβαια το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Ωστόσο διάφορα ζητήματα έχουμε ήδη προγραμματίσει να θέσουμε. Είμαι σίγουρος ότι στη Διυπουργική η Υπουργή, η Επίτροπος Μάλστρομ θα είναι σε θέση να υιοθετήσουν το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του συστήματος επίλυσης συγκρούσεων που προβλέπει η Συμφωνία. Θα προσπαθήσουμε επίσης να έχουμε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και την παρακολούθηση της Συμφωνίας Εταιρική Σχέσης. Όπως γνωρίζετε κύριε Σούστα, έχουμε προσπαθήσει να πείσουμε τους εταίρους μας στην Νότια Αφρική ότι χρειάζεται να εμπλέκεται η κοινωνία των πολιτών στον έλεγχο και στην παρακολούθηση της συμφωνίας και ότι αυτό θα πρέπει να καταγραφεί και τυπικά, να ε, θεσμοποιηθεί. Δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει σε αυτό, δεν έχουν δεχτεί αυτή την πρόταση. Συνεχίζουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης έχουμε προτείνει έναν μηχανισμό για την αποκοινού παρακολούθηση του, της συμφωνίας. Συνεχίζονται λοιπόν οι συζητήσεις και θα συνεχιστούν και στις 6 Νοεμβρίου, εν μάλλον τη συνάντηση της 6 Νοεμβρίου στο Ιωάννεσπρο. Σας ευχαριστώ. Την τελευταία, τον τελευταίο λόγο Γενική Εισηγήτρια, κυρία Χίρης. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Κομισιόν και τον ε, πρέσβη και την ε, ομάδα του. Όπως είπε και ο συνάδελφος, πραγματικά είναι σημαντικό κυρίως να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε όλα αυτά τα θέματα που άπτονται του διαλόγου με την Κοινότητα των πολιτών που είναι μια πολύ σημαντική πτυχή για εμάς και πολύ σωστά υπόθηκε ότι υπερβαίνει τις καθαρά οικονομικές πτυχές της συμφωνίας. Είναι μια πρόκληση, όμως νομίζω ότι είμαστε γενικά στο σωστό δρόμο και θα πρέπει να δούμε ε, και τι θα προκύψει στη συνέχεια και θα περιμένω να δω ε, πώς θα το παρακολουθήσει το θέμα η αν θα μας στηρεί ενήμερος, κάτι που το ελπίζω, γιατί οι συνάδελφοί μου και εγώ θέλουμε να έχουμε στοιχεία και από τα στατιστικά και από την ε, Σύνοδο Κορυφής. Θέλουμε λοιπόν να τηρούμε θα ενήμερη. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το σημείο της μερίσιας διάταξης. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του όλους ιδιαίτερος ε, τον πρέσβη της Δημοκρατίας της ε, Νοτιοαφρικής. Ε, να ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας τους που ήταν εδώ και για την ανταλλαγή απόψεων. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε αμέσως στο επόμενο σημείο, υπαριθμόν 12, της ημερήσιας διάταξης. Κατάσταση συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Ήδη είναι εδώ ο εισηγητής μας, ε, ο κύριος Αλαφράνκα. Και θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης σε ό,τι αφορά την κατάσταση συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, Αυκό είναι καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως εξηγήσατε, επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου συνεισφέρει σε αυτή την έκθεση για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι προφανές ότι η πολιτική για το εμπόριο είναι μία από τις θεμελιώδες, τα στοιχεία ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε κάποιες σκέψεις δηλαδή για το πώς εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί αυτή η πολιτική που είναι μία από τις ε, ιδρυτικέ πολιτικές τη ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης και θα συνεχίσει να έχει μεγάλη σημασία τα επόμενα χρόνια. Η πολιτική για την ανάπτυξη γενικά. Είναι ε, κάτι το οποίο μπορεί να φέρει πρόοδο, να φέρει ειρήνη. Γι' αυτό θα πρέπει να διατυπώσουμε ορισμένες βασικές αρχές που να μας κατευθύνουν στο μέλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η έκθεση την οποία υποβάλλω στα μέλη. Να προτείνουμε δηλαδή με ποιον τρόπο η Ευρώπη θα είναι ηγετική, σε ηγετική θέση έτσι ώστε να προωθήσει ένα σύστημα δίκαιο για το διεθνές εμπόριο που να βασίζεται σε διεθνεί συμφωνίες έτσι ώστε οι κανόνες να, να εφαρμόζονται και έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να ανταγωνίζονται, να δραστηριοποιούνται και διεθνούς με ξεκάθαρους κανόνες. Αυτό είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε συμφωνίες διεθνού εμπορίου με Πρωτογνωσιακό καθεστώτα. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Βεβαίως θα πρέπει να θέσουμε σε προτεραιότητα εκείνες τις χώρες με τι οποίε επιθυμούμε να έχουμε διμερείς συμφωνίες, και βεβαίω να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει στο πλαίσιο του ΠΟΕ και να συνεισφέρουμε στη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός. Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, όπου βλέπουμε να επανέρχεται ο προστατευτισμός και να υιοθετούνται μέτρα τα οποία είναι ενάντια στα συμφέροντές μας και στις αρχές μας, θα πρέπει να το προσπαθήσουμε αυτό. Από εδώ και πέρα, μιλώντας για τα ζητήματα που είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρεμβαίνουμε και θα θέλαμε να ζητήσουμε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτέ τι διαδικασίε να συμμετέχει πλήρω. Αποτελεί εξάλλου και μία μέρο τη συμφωνία δια... μεταξύ των θεσμικών οργάνων και είναι και κάτι το οποίο ανέφερε και ο Προεδρο τη Επιτροπή στην πρόσφατη ομιλία του για το μέλλον τη Ευρώπη και είναι και κάτι το οποίο έχει αποδείξει την αξία του. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε και την εμπειρία τη Επιτροπής της κοινοβουλευτική για το Διεθνές Εμπόριο, αλλά και άλλες δυνάμεις και άλλους ειδικού για το θέμα, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει καλύτερα στι διαπραγματευτικές διαδικασίε. Κάτι ακόμα που θεωρώ σημαντικό είναι η φορά που κάνουμε στο ότι η προθεσμία και το η ταχύτητα με την οποία γίνονται αυτέ οι διαπραγματεύσει πρέπει να είναι πιο λογικέ, γιατί χάνουμε ευκαιρίε. Σε πολλέ περιπτώσει φτάνουμε τελευταίοι. Καθυστερούμε. Δεν μιλώ μόνο για το ζήτημα της επικύρωσης, ακόμα και πρόσφατο παράδειγμα έχουμε στην ανανέωση της συμφωνίας με το Μεξικό φαίνεται ότι η ανανέωση της συμφωνίας με το Μεξικό θα πάρει περισσότερο χρόνο από ό,τι πήρε η πρώτη σύναψη της συμφωνίας. Πέρα από αυτό, θα πρέπει να δούμε το ζήτημα του ψηφιακού εμπορίου, της κοινοτομίας, της ψηφιοποίησης και να το εντάξουμε αυτό στις ε, διμερείς και πολυμερείς μας διαπραγματεύσεις. και να αξιοποιήσουμε επίσης το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχουν αρνητικές συνέπειες. Συμφωνούμε όλοι νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι χρειάζεται συντονισμός στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στον τομέα Τη εμπορικής πολιτική με τις πρωτοβουλίε που αναλαμβάνουμε στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, καθώ επίσης και στον τομέα της οικονομικής πολιτικής. Ιδίω όταν εξυγχρονίζονται τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και επίσης το ίδιο συμβαίνει και με την πολιτική που έχουμε στον τομέα της ε, ανάπτυξη, τη αναπτυξιακή βοήθεια, μάλλον. Κλείνοντα θα έλεγα ότι δεν μπορούμε ακόμα να γνωρίζουμε τελικά προς τα πού θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως σε κάθε περίπτωση, θα, μετά το Brexit, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να έχουμε το ελάχιστες δυσμενείς επιπτώσεις. Πιστεύω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να κάνει μια καλύτερη δημοσιοποίηση, παρουσίαση των θετικών στοιχείων που έχουν οι εμπορικές μας πολιτικέ για την αύξηση του καθαριστών χωρίου προϊόντος, για τη δημιουργία θέσεων εργασία. και να δείξει πώς επιχειρήσεις και πώς οι πολίτες μας τελικά μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα αυτές τις ευκαιρίες που οι συμφωνίες, οι διεθνείς συμφωνίες εμπορίου μας δίνουν. Κλείνω Λέγοντα ότι βεβαίω προσβλέπω στη συνεργασία με του ε, συναδέλφου και τα σχόλια και τι παρατηρήσει που θα μου υποβάλλουν επί τη γνωμοδότησής μου. Βεβαίω γνωρίζετε ότι υπάρχουν συνηθισμένοι περιορισμοί χώρου, ε, της έκτασης της έκθεσης δηλαδή, που υποβάλλουμε. Αλλά βεβαίω ε, είμαι σίγουρο ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε και άλλε στοιχεία σε αυτήν. Σα ευχαριστώ πολύ. Εμεί ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Καλώ ήρθατε κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να πάρετε τη, το, την Προεδρία. Όχι. Να ολοκληρώσω και σα δώσω και τα άλλη μετά τότε. Δυστυχώ ε, δεν είναι εδώ άλλο συζητητή από την ΑΦΚΟ. Επειδή και εκεί συζητείτε το ζήτημα, οπότε θα περάσω στου κοιόδη συζητητέ αυτής αμέσω. Ε, Αρχέ γενομένε από τη Μαρία Ρενά, από Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ απόλυτα ω προ το ότι η εμπορική πολιτική τελικά, επιτέλους θα έλεγα, έγινε μια πραγματική πολιτική. Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια εμπορική τεχνική, τεχνική προσέγγιση. Το εμπορίο έχουμε περάσει την πολιτική προσέγγιση του εμπορίου και πολύ με ικανοποιεί αυτό που είπε ο κύριο Αλαφράγκα, ότι η εμπορική πολιτική είναι ένα πραγματικό εργαλείο στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει βέβαια να ευνοεί αυτό το εργαλείο την ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όμω ότι είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη, όπω εμεί την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια δίκαιη ανάπτυξη του Ευρωπαίου. Υπάρχει δηλαδή επιστροφή. Ε, υπάρχει όφελος για όλο τον ευρωπαϊκό πληθυσμό και χαίρομαι που ο κύριος Σαλαφράγκα προωθεί και προβάλλει το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που μπορεί να παίξει έναν ρόλο αλληλεγγύης, παροχής αλληλεγγύης για τα άτομα που δεν είναι ευνοημένοι από την εμπορική πολιτική, που δεν είναι αυτοί αποδέκτες κατά αναγκευτής της πολιτικής, αλλά θέλουμε να υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση και απέναντι στους εμπορικούς μας Θα πρέπει η εμπορική πολιτική να ασκείται σε ένα πλαίσιο που θα έχουμε κατά νου τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα αφορά τα κλιματικά ζητήματα. Θα πρέπει να λαμβάνεται η διάσταση του κλίματος στην εμπορική πολιτική για να αποφύγουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη και να πετύχουμε τους στόχους της ε, COP21. Φυσικά και θέλουμε να προωθήσουμε το πολυμερές σύστημα που περνάει δύσκολους καιρούς σήμερα, αλλά είναι ένα σημαντικό εργαλείο αυτή η συμφωνία. Πρέπει να μιλήσουμε για τρία σημεία σε ό,τι αφορά αυτή την εμπορική πολιτική. Τι αξίες μεταφέρουμε μέσω αυτής της εμπορικής πολιτικής. Για παράδειγμα, μιλήσαμε ε, διαμακρών για τη, τα δικαιώματα στην εργασία, τι συμβάσει τη ε, ΔΟΕ και το συζητούμε σε εμπορικές μα συμφωνίες. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό για εμάς, είναι η διαφάνεια αυτών των εμπορικών πολιτικών που ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ε, τις βλέπει με πολύ κριτικό πνεύμα, δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι γίνεται. Η διαφάνεια λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό και το τρίτο είναι η πανεξισορρόπηση των εμπορικών συμφωνιών. Σήμερα είναι όλο και πιο ευρειε αυτές οι συμφωνίες, δεν περιορίζονται στους δασμούς. Είναι σημαντικό λοιπόν οι εμπορικέ συμφωνίε αυτέ, επειδή μιλάμε για ρυθμιστική συνεργασία, κανονιστική συνεργασία, να μιλάμε και για κοινωνική, περιβαλλοντική αλλά και φορολογική συνεργασία στο πλαίσιο των συμφωνίων αυτών. Και νομίζω ότι θα καταθέσουμε σχετικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. ECR. Ο Σάντρε Λούνες δεν είναι εδώ. Από την Άλντε η κυρία Λαλόντ δεν είναι εδώ. Από τις πράσινους ο κύριος Μπούχνερ δεν είναι εδώ. Είναι όμως εδώ ο κύριος Χέλμουτ Σόλτς από την ΚΟΕ και έχει και το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη πρόκληση ε, να συζητήσουμε το μέλλον της ε, κατάστασης ένωσης ε, και το έχει αναλάβει η Επιτροπή Συνταγματικών. Υποθέσω να άξω πολύ προσεκτικά την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει στη γνωμοδότησή του ο συντάκτης μας, ο κ. Σαλαφράγκα. επειδή είμαι στην Επιτροπή Συνταγματικών και γνωρίζω λίγο πολύ αυτή τη συζήτηση, Το θέμα είναι να συνεισφέρουμε με κάποιο τρόπο για να έχει ένα μέλλον η κοινωνική δημοκρατική Ευρώπη. Και επομένως πρέπει να επηρεάσουμε και την εμπορική πολιτική. Άρα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα σε σχέση με τις προτάσεις ε, του κυρίου Σαλαφράγκα. Θα συζητήσουμε για συνέκταση για την παγκοσμιοποίηση. Τέτοια πράγματα πρέπει να γίνουν. Τα είπαμε και σε άλλε εκθέσει. Σε σχέση και με τον ΠΟΕ, για παράδειγμα. Έχουμε τις, ε, τα benchmark. Ε, πρέπει να τα αναφέρουμε ξεκάθαρα για την εμπορική Πρέπει να εφαρμοστούν, πρέπει να υλοποιηθούν και σε επίπεδο κρατών μελών της Ένωσης. Ε, έχουμε συζητήσει και ξέρουμε και τι έγινε με την TTIP, τη ΣΕΤΑ ε, και οι πολίτες της Ευρώπης ενδιαφέρονται και θέλουν να υπάρχει μια εμπορική πολιτική που να εκπροσωπεί και να υπηρετεί τα συμφέροντά τους. Ε, συμφωνώ για τη διαφάνεια, είναι πάρα πολύ σημαντική και η διαφάνεια αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Οι στόχοι της βιωσιμότητας πρέπει να είναι αυτό το σημείο αναφορά benchmark, αν μπορώ να το πω έτσι, ε, για, την, ε, για το μέλλον της Ευρώπης. Και ένα άλλο θέμα και ένα άλλο ερώτημα είναι συνεργασία μας ε, στο επίπεδο της εμπορικής πολιτικής, πώς θα την αναπτύξουμε ώστε να είναι προς όφελος των μικρομεσών επιχειρήσεων, των μικρομεσών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν μια τύχη, μια ευκαιρία στην ε, παγκόσμια αγορά, να μην αποδοπατηθούν, μπορούν να έχουν ε, πρόσβαση και να έχουν πρόσβαση και σε άλλες αγορές, σε άλλα μέρη του κόσμου. Είναι και αυτά θέματα. Έχουμε νέες επίσης εξελίξεις, έχουμε την ψηφιοποίηση κτλ. κτλ. Πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα και η Επιτροπή υποθέσεων. Πρέπει να τα λάβει αυτά υπόψη της όταν ε, θα συζητήσει ε, το μέλλον της έξευσης της Ευρώπης και έχουμε τα βιομηχανικά επίσης ζητήματα πέραν των πολιτικών κοινωνικών που πολύ ενδιαφέρον. Εγώ αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα από κοινού να ακολουθήσουμε και να σκεφτούμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να δομήσουμε έτσι αυτή την γνωμοδότηση και να πω και κάτι ακόμη. Νωρίσιμα το πρωί μιλήσαμε για την ε, συμφωνία με την Ιαπωνία. Πολλά θα ξέρω. το αν είμαστε ανοιχτοί και από την ανάπτυξη των άλλων περιοχών και να δούμε κατά πόσον εκεί θα αναπτυχθεί μια βιώσιμη ε, πολιτική, εμπορική βιομηχανία κτλ. ή αν θα πάνε ως μοναχικοί καβαλάριδες ε, οι άλλες χώρες. Και ε, ξέρετε ότι δεν είναι μόνο η Ιαπωνία, έχουμε και άλλες. Ε, έχουμε τη σχέση με τις χώρες Αφρικής, ε, με τη Λατινική Αμερική. Είμαστε και εμείς υπεύθυνοι. Πρέπει να χαρακτηρίζεται η πολιτική μας από υπευθυνότητα για να προχωρήσουμε. Και βεβαίω και ολοκληρώνοντα να πω ότι περιμένω τη συνεργασία μα με τον εισηγητή και του άλλου και και ότι φυσικά θα καταθέσουμε τροπολογίε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ακόμα δύο εγγεγραμμένου στον κατάλογό μου, ο κύριο Στάκμελ και η, Μακουλάδα Ροντρίγε Πινιέρο. Ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Ωραία, επομένω ολοκληρώνεται ο κατάλογο και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντάχνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, θα, ήθελα να ζητήσω κάποιε διευκρινήσει ε, ε, από την ΑΦΚΟ, όχι από εμά πάντως, αποτελεί το μέλλον της Ευρώπης. Και το περισσότερο κομμάτι της, του κειμένου αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο Ευρώπη και δεν είναι, ε, τι να σας πω, σημείο έτσι, ακαδημαϊκής σκέψης. Είναι μια πραγματικότητα ε, και μετά τον Μάρτιο η πραγματικότητα αυτή θα είναι μπροστά μας. Ε, επίσης όλες αυτές ε, οι επιτροπές έχουν πολλούς υπαλλήλους. Άρα Πολλοί είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι θα μπορούσαν πρώτον να τα σκεφτούν, αλλά εν πάση περιπτώσει εκ των υστέρων να τα διορθώσουν. Στο σημείο 6 ε, αναφέρεται <clears throat> στην διευκόλυνση την πρόσβαση ε, προς την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή τι ε, στην ουσία εδώ αναφέρεται τρομερή αύξηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης αυτό σημαίνει, εάν ζητούμε τέτοια προσβασιμότητα, τότε θα υπάρχουν οπωσδήποτε περισσότερες αιτήσει και άρα περισσότερα χρήματα. Ε, θα ήθελα απλώς διευκρίνηση και εδώ, όπως και στο πρώτο σημείο. Τρίτον, αλλά πολύ σαφές ε, εδώ, αναφέρεται ότι το εμπόριο θα χρησιμοποιηθεί σαν ε, ε, εργαλείο, σαν όπλο για την ε, εμπορική πολιτική. Επανειλημμένα έχω αναφερθεί στην πολιτικοποίηση του εμπορίου. Και μάλιστα ο πρέσβης της Αργεντινής που μίλησε προηγουμένως ε, είπε ότι το εμπόριο, κυρίως δε το ελεύθερο εμπόριο ε, διευκολύνει την ε, ανάπτυξη. Αλλά όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια υπερδομή από, δομέ, από ε, θέσφατα, υποθέσεις εργασίας και λοιπά και αξίες και τιμές, τότε οπωσδήποτε αυτό θα έχει το περίεργο δύσκολο οικοδόμημα, θα έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερο εμπόριο. Το σημαντικό είναι βέβαια ε, να ε, προωθήσουμε την ευημερία. Αλλά η χρήση της εμπορικής πολιτικής σαν ένα εργαλείο της εξωτερικής ε, ε πολιτικής είναι μία άποψη. Απλώς θα ήθελα εγώ να χτυπήσω ένα καμπανάκι όσον αφορά τις επιπτώσεις μιας τέτοιας τάσης και μιας τέτοιας πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ η Μακουλάδα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε και τον εισηγητή ε, για την γνωμοδότηση την οποία μας ε, παρουσίασε. Πιστεύω ότι ε, σε γενικές γραμμές μπορούμε να δεχτούμε τις αρχές. Τώρα το τι μέλη γενέστε είναι άλλο και επί του πρακτέου δεν μπορούμε να πούμε και πολλά γιατί εδώ υπάρχει ένα περιθώριο, μάλλον ένας περιορισμός μήκους. Υπάρχει κι άλλο ένα ε, θέμα το οποίο θα ήθελα ε, να... Μάλλον όχι, τέσσερα σημεία θα ήθελα να ε, θίξω. Όταν λέμε ότι πρέπει να είναι συμπεριληπτική η εμπορική πολιτική και ότι θα πρέπει να οδηγήσει προς πιο δίκαιη παγκοσμιοποίηση, εγώ πάντα σκέφτομαι το 50% του κόσμου που δεν ε, μπαίνει στις εμπορικές συμφωνίες και εν πάση περιπτώσει ε, επιμένω ότι θα πρέπει να ε, συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου σε όλες αυτές τις, σε όλες αυτές συμφωνίες και άλλωστε έχει υπάρξει και σχετική συντριπτική πλειοψηφία κατά την έννοια αυτή και στην Ίντα και στη φάμα. Προηγουμένως συζητήσαμε για την Ιαπωνία και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν ε, ε, ε, πρόσβαση σε όλα αυτά. Τρίτον, στην πολιτική γενικά, αλλά και στην εμπορική πολιτική, ο κίνδυνος που διατρέχουμε είναι η διατάραξη της παγκόσμιας τάξης και θέλουμε να αποφύγουμε να επαναληφθούν ε, ας πούμε οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε πολυμέρεια και η παγκόσμιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου είναι αυτός που καλύτερα ασχολείται με τις πολυμερείς σχέσεις, άρα θα πρέπει να του, τον αναζωογονήσουμε. Τέλος, το είπε και η Μαρία Αρένα κάποια στιγμή σε σχέση με την φορολογική πολιτική και την δυνατότητα ε, να χρησιμοποιηθούν οι εμπορικές συμφωνίες για αυτήν την διεθνή ε, συμφωνία με οδηγούν στο θέμα της διαφθοράς ε, και συγκεκριμένα της μάχης κατά της διαφθοράς. Εάν δεν αποτελεί σημείο εστίασης με τις χώρες με τις οποίες συναλλασσόμεθα, Πιστεύω ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ε, την, ε, μια ε, πραγματικά φιλόδοξη και θαραλέα εμπορική πολιτική. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Λούκα Δικάρλη από την DigiTrade. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή για τις θέσεις του. Είναι δύσκολο σίγουρα να πρέπει να συντάξετε μια τόσο ε, σύντομη σε έκταση, έκθεση για το μέλλον της Ευρώπης. Το είδαμε αυτό και σε προηγούμενε γνωμοδοτήσει. Υπάρχουν γνωμοδοτήσει ε, για το Ταμείο για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων τη Παγκοσμιοποίηση και άλλε με τι οποίε συμφωνώ. Συμφωνώ με πολλέ από τι παρατηρήσει που έγιναν. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι όσον αφορά αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής. Όταν λέτε ότι θα πρέπει να διευκολυθεί η πρόσβαση σε αυτό έτσι ώστε να προκατα... προλαμβάνουμε τις επιπτώσεις, Βεβαίως εμείς θα θέλαμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στο ταμείο αυτό. Έχουμε προτείνει για παράδειγμα αύξηση ε, του συνολικού προπολογισμού του 15%. Έχουμε προτείνει μείωση των κατοφλίων, αλλά το EGF, αυτό το ταμείο, από τη φύση του επεμβαίνει εκ των υστέρων, όταν έχουν πληγεί οι άνθρωποι. Κάνουμε κάποια προβλέψεις, κάποιες, αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Υπάρχουν άλλα εργαλεία, ε, τα κοινωνικά ταμεία, τα διαρθρωτικά ταμεία, τα, ταμεία, τα περιφερειακά, ε, και το ΕΦΣΥ που μπορούν να συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μάλλον, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προλαμβάνει κανεί τι καταστάσει. Αυτό από την πλευρά μου ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Σαλαφράγκα, τον εισηγητή μα, λέει ο πρόεδρο. Κύριε Σαλαφράγκα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και του συναδέλφου και τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι παρατηρήσει του, που σίγουρα θα εμπλουτίσουν την γνωμοδότησή μου. Θα ήθελα να πω στην κυρία Αρένα μιλάτε για ένα εμπόριο το οποίο βοηθάει την ανάπτυξη, που αυτό να γίνεται με τρόπο δίκαιο. Όταν μιλούμε για δικαιοσύνη, δεν μιλούμε μόνο για δικαιοσύνη μεταξύ των μερών που συμμετέχουν, αλλά μιας και μιλούμε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλούμε επίσης και για ηθικές αξίες, τις οποίες θα πρέπει να δεσμεύουν και τα δύο μέρη. Είμαστε υπέρ του ανοιχτού εμπορίου με αηφορία και με βιωσιμότητα, αυτό το προωθούμε και θα θέλαμε να σκεφτούν οι αντίστοιχες συμφωνίες. Θα πρέπει όμως να αντιτυπώται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχουμε και αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε τελικά το εμπόριο, η αύξηση του εμπορίου να βοηθάει και τις επιχειρήσεις μας και τους πολίτες. Αναφερθήκατε επίσης στην COP21 και στην κλιματική αλλαγή. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό πράγματι να αναφερθεί και αυτό αποτελεί εξάλλου και μέρος των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, είναι γνωστό. Θα το προσθέσω λοιπόν, θα προσθέσω μια σχετική παραπομπή στην εκθεσή μου. Κατά τα άλλα, το ζήτημα της διαφάνειας, πιστεύω ότι και αυτό μπορεί να ενταχθεί στους στόχους που προσπαθούμε να πετύχουμε. Και όσον αφορά τώρα τις αρμοδιότητες και τη σχέση με τον Παγκόσμιο Οργάνωση Εργασίας ε, αποτελεί και αυτό μία από τις προτεραιότητές μας όταν αναλαμβάνουμε τέτοιες συμφωνίες. Τους σκιώδες του ECR και την ALDE δεν ήταν εδώ. Άκουσα τις παρατηρήσεις του κ. Σόλτς από την ΚΟΕ. Μου φαίνεται πολύ σημαντικό αυτό που είπε για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την, την συνεισφορά, τη βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Βεβαίω να κάνουμε μια αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ πιστεύω ότι αν και οι μικρομεσαίες έχουν τεράστια σημασία αυτές οι επιχειρήσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Άκουσα με προσοχή την παρέμβαση του κ. αλλά αυτά που λέει είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Και θα προσπαθήσω, προσπαθώ να βρω κάτι με το οποίο να μπορεί να επιτύχουμε σύνθεση των απόψεων, με θετικό τρόπο. Ε, αυτό που μας λέει ο κύριος Ντόρτμοντ είναι ότι εμείς που υποβάλλουμε μια γνωμοδότηση προς την υπόθεση, ε, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, εκείνη είναι που εξετάζει το μέλλον της Ευρώπης, βεβαίως έχετε δίκιο ότι το, η Ευρώπη είναι μια έννοια η οποία προϋπάρχει της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αλλά από τη ε, διαδικασία που έχει την επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή είμαστε περιορισμένοι σε αυτό που μου ζητάτε. Τώρα, σε αυτό που λέτε για το, τη ρύθμιση του παγκοσμίου εμπορίου, η διαφορά μας με άλλες μεγάλες δυνάμεις είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιωμένη σε αξίες, σε αρχές. Και για μας αυτές οι αξίες και αρχές είναι σημαντικές και ζητούμε την αμοιβαία εφαρμογή τους δεν σημαίνει αυτό ότι δίνουμε μαθήματα στις άλλες χώρες, αλλά ζητούμε εφαρμογή και από τα δύο μέρη, αμοιβαίω. Και επομένω, οι εμπορικέ μα συμφωνίες ε, θεμελιώνονται στη βάση αυτών των αρχών και αξιών. Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι υπερβολικό ε, και πράγματι πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται με με προσοχή, χωρί να, να, να, δημιουργεί υπερβολικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε αυτό μόνο συμφωνώ με τον κύριο Ντόρκμουντ. Γνωρίζουμε επίση ότι εξαιτία του ελεύθερου εμπορίου πολλέ φορέ δημιουργούνται ασύμετροι Θα μπορούσε να το πει κανεί αυτό για τη συμφωνία με την Ιαπωνία όταν ε, γνωρίζουμε το μέγεθος αυτή της οικονομίας 30% ε, και Όμω όταν συζητούμε συμφωνίε, για παράδειγμα με την Κεντρική Αμερική, με την Χιλή που το μέγεθος της οικονομίας τους είναι πολύ μικρότερο από εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωση και έχουν πολύ διαφορετικές πολιτικές, ε, Πολιτικά έχουμε εναντί του. ε, είναι λογικό να ζητάει κανείς μεγαλύτερη προσοχή όταν συνάπτουμε συμφωνίες με τέτοιες χώρες, να προσέχουμε τι επιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν αυτές τις συμφωνίες για πολλούς ανθρώπους. Μιλούμε για την παγκοσμιοποίηση και την ανάπτυξη με ανθρώπινο πρόσωπο που θα προωθεί την αξιοπρέπεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό να αποφύγουμε την όποια υποστοχώρηση. Προσπάθησα να το διατυπώσω αυτό διπλωματικά, λέγοντας ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση. Δεν σημαίνει αυτό, κύριε Ντόρτμοντ, ότι ζητούμε περισσότερα χρήματα, γιατί είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να περιοριστούμε στο πλαίσιο του τρέχοντος πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και δεν είναι τώρα η ώρα. Κάποια στιγμή, όταν συζητηθεί το πουδο που θα στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ο καθένα θα εκφράσει τη θέση του από αυτού. Ε, έχουμε το προενταξιακό εργαλείο, 14 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιούνται. όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα προ τι εμπορικέ συμφωνίε. Όμω εδώ συζητούμε πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει τι τις ε, εμπορικέ τη συμφωνίε, έτσι ώστε αυτέ να έχουν θετικό αντίκτυπο οι ίδιε και επίση τι άλλα εργαλεία μπορεί να αξιοποιήσει έτσι ώστε να αντισταθμίσει πιθανέ αρνητικέ επιπτώσει των συμφωνιών. με τρίτε χώρες. Αν κάνει κανείς μια ανάλυση των αποτελεσμάτων, είναι ξεκάθαρο ότι οι συμφωνίες αυτές έχουν συνεισφέρει στην αύξηση του ΑΕΠ, στη μείωση των ανισοτήτων, αύξηση των εξαγωγών, τα ξέρετε αυτά. Και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους, όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα αυτούς που το χρειάζονται. Κύριε Πινιέρο, Πινιέρο Συμφωνώ μαζί σας πλήρως. Θα βρω, θα συζητήσουμε και μαζί αν θέλετε πώ ακριβώς να το εντάξουμε στο νομοδότησή σα Θα πρέπει να εντάξουμε και το ζήτημα του φύλου. Ε, μίλησε ήδη για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θα πρέπει να βρούμε ίσω μια διατύπωση που αναφέρει πόσο σημαντικές είναι για την ε, οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωση αυτέ οι επιχειρήσει. και νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Πράγματι, η πολυμερής προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις είναι ένας κίνδυνος που θα πρέπει να αποσοβήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα αυτό. Έχουμε συνεισφέρει στη δημιουργία ενός διεθνού συστήματο που με όλα του τα προβλήματα έχει λειτουργήσει. Και τώρα περνάμε μια δύσκολη περίοδο ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ποια είναι τα όρια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην πολιτική μας ολοκλήρωση. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε, να, να, να ε, πούμε με μεταβεβαιότητα στους πολίτες μας ότι κάτι το οποίο λειτουργεί και το οποίο το είχαμε ήδη από το ακούσει από τον Οκτώβριο του 2014 όταν ανέλαβε η νέα επιτροπή, το είχε πει ο κ. Γιούγκερ, ότι αυτή η επιτροπή θα είναι η επιτροπή της τελευταίας ευκαιρίας Πράγματι λοιπόν έχουμε πολλές δυσκολίες, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η εμπορική πολιτική λειτουργήσε προς όφελος των πολιτών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε αντικρουόμενες απόψεις, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τις συνθέσουμε, έτσι ώστε η πολιτική αυτή να λειτουργήσει προς όφελος των επιχειρήσεων μας, προς των πολιτών, προς όφελος των εργαζομένων, προς όφελος όλων. Ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά τους σε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση η οποία θα υπερψηφιστεί από την Επιτροπή μας με μεγάλη πλειοψηφία και η οποία θα αντικατοπτρίζει όλες τις θέσεις και τις απόψεις που, έχουν, που έχετε εκφράσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Uh, we Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Άψογοι είμαστε ε, στο χρόνο μας. Ε, έχουμε, είμαστε πέντε λεπτά, ε, έχουμε κερδίσει πέντε λεπτά. Να σας υπενθυμίσω ότι ε, η, αυτή την Παρασκευή το μεσημέρι, δηλαδή 12 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι λίγη η προθεσμία υποβολής τροπολογιών και στις 5 Νοεμβρίου θα συζητηθεί στην Επιτροπή μας αυτά και θα δώσω το λόγο στον, θα δώσω την Προεδρία, θα την παραδώσω στον Πρόεδρο. So, thanks a lot, Mr. Vice Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε που προεδρεύσατε όσο έλειπα. Ζητώ συγγνώμη αλλά ήμουνα σε μια πολύ σοβαρή συζήτηση, ε, συνάντηση με την European Enterprise ε, στο ημικύκλιο και συζήτηση με την ε, κυρία Μάλστρομ. Θα πάμε τώρα στο σημείο 13. Είναι ένα θέμα που αφορά την Κίνα. Ο κύριος Βίνκλερ είναι αυτός που τα ξέρει όλα για την Κίνα και θα μας τα πει αμέσω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα ε, για το οποίο είχαμε ανταλλαγή ε, επαφών, σχετικά, ε, επιστολών συγγνώμη, σχετικά με τα κοτόπουλα. Είναι τεχνικό ζήτημα, όπως σας είπα και προηγουμένως. Η πρόταση που βρίσκεται ενώπιόν μας ε, ε λέει ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε ε, να υλοποιηθεί η απόφαση ε, της 17 Απριλίου του 2017 του ΠΟΕ που αφορά ακριβώς σημεία δασμολογικές παραχωρήσεις για προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών. Είχε απαγορευτεί η εισαγωγή ε, ε, προϊόντων με βάση κρέας πουλερικών ε, λόγω με βάση της απόφασης αυτής και λόγω προβλημάτων ζωονόσων. Το πάνελ του ε, ΠΟΕ του Ιουλίου 15 συστάθηκε για το θέμα αυτό και έλαβε υπόψη ε, πολλά θέματα, δύο ε, εκ των οποίων ήταν οι δασμολογικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί Δύο έγιναν ε, δεκτές και άλλες ε, οκτώ ε, απερίφθησαν σε αυτήν την εξέταση της διαφοράς. Την 16η Μαΐου του 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφόρησε το Σώμα Επίλυσης Διαφορών ότι θα υλοποιήσει τις συστάσεις που είχε λάβει και ζήτησε εύλογο χρονικό διάστημα για την περίοδο αυτή εφαρμογής που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017. Η Κομισιόν διαπραγματεύτηκε συμφωνία με την Κίνα έτσι ώστε να βρεθεί αποδεκτή λύση. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να σας τα πω όλα. Στην αιτιολογική επεξήγηση τα βρίσκεται όλα. Το θέμα είναι ότι τώρα ε, έχουμε ε, λίγο χρόνο στη διάθεσή μας ε, και πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία έτσι ώστε να αναφερθούμε στο πάνελ του ΠΟΕ. Η απόφαση της ε, Κομισιόν, κατά την άποψή μου, είναι σωστή. Τα μέτρα και ο τρόπος με τον οποίο ε, ε, αντιμετώπισε το θέμα είναι ορθός. Έχει προβλεφθεί τέλος του μήνα να υπογραφεί η σχετική συμφωνία στην Γενέβη. Ελπίζουμε δηλαδή αυτό να καταστεί δυνατόν. Θεωρούμε ότι μπορούμε να δώσουμε την σύμφωνη γνώμη μας στην συμφωνία αυτή. Πάντως, όπως πάντα και ως εισηγητής, ε, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, συμφωνήσουμε με αυτήν την θέση όσον αφορά τον πόλεμο. <laughs> Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Εξαιρετικά. Έχουμε σκιώδη εδώ. Μη μου πεις, λέει ο πρόεδρος. Helmut Σόλτ. Πολύ σύντομα θα το πω. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να συνεχίσετε να πηγαίνετε ε, σε κινέζικα εστιατόρια και να παίρνετε για πιάτο, ας πούμε, για να φάτε πια, πάπια Πεκίνου, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να καλωσορίσετε αυτήν την θέση και αυτήν την συμφωνία. So, even e. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι συμφωνεί ακόμα και η Γκουε e με το κείμενό μου. Wow, λέει ο μιλητής. Ε, η Λουσία Κόσε Γουγανόβα από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να σπαταλήσω το χρόνο σας, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον ε, εισηγητή κύριο Βίνκλερ ε, ε, Λούλου για, το, για την τοποθέτησή του μονάχα να υπογραμμίσω δύο σημεία τα οποία τα αναφέρατε κι εσείς άλλωστε. Πρόκειται για συμφωνία αμοιβαία όσον αφορά, την, ε, όσον αφορά υλοποίηση αποφάσεων του πάνελ επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Ε, είμαστε και ε, μας ζητήθηκε να συμμορφωθούμε με τα ευρήματα ε, σε εύλογο χρονικό διάστημα που είναι 15 μήνες ε, και αυτοί ε, οι μήνες ολοκληρώθηκαν τον του 17 Δεύτερον, τα ευρήματα του πάνελ ήταν θετικά και καθυσυχαστικά, κυρίως όσον αφορά την συστηματική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις άρθρο 28. Πάρα πολύ ωραία. Θέλει ο εισηγητής να πει κάτι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στον εκπρόσωπο της Γκουε για την υποστήριξή του. Χέλμουτ, έχουμε πάει τόσες φορές μαζί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ε, που ε, καταλαβαίνω ε, ότι το, το κείμενο αυτό δεν το έγραψα γιατί μ' αρέσει η Παπια Πεκίνου, αλλά γιατί έχω παρακολουθήσει από κοντά το πλαίσιο του ΠΟΕ. 12 ε, Οκτωβρίου λίγη η προθεσμία υποβολής τροπολογιών στις 12 ακριβώς. Ε, βέβαια δεν είναι πολύ χρόνος, ίσως δεν υποβληθούν τροπολογίες, ωστόσο κανείς δεν ξέρει. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα κάνουμε μία μικρή διακοπή μέχρι τις 4.30 αλλά ίσως καλύτερα να έρθετε 4 και 25. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε 4 και μισή.

Ευχαριστώ. So, uh, and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, αγαπητοί φίλοι, θα ξεκινήσουμε τώρα την ε, ακρόασή μας σχετικά με τη Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ. Χαίρομαι γιατί διαπιστώνω ότι έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ακρόαση. Και νομίζω ότι έγκαιρα ε, οργανώνεται αυτή η συνεδρίαση. Έχουμε μακρά ιστορία όσον αφορά αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα έδειξε μεγάλη, πολύ καλή διάθεση ε, και εν τέλει έχουμε δύο συμφωνίες, ε, μία για την προστασία των επενδύσεων και μία για το εμπόριο. Αυτό γιατί υπάρχει ειδικό σύστημα προστασίας των επενδύσεων ε, και πρόκειται επίσης για ζητήματα τα οποία αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Έχουμε τώρα λοιπόν μια φιλόδοξη συμφωνία, εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός ε, και αυτήν την αναπτυσσόμενη χώρα που νομίζω ότι αποτελεί υπόδειγμα καλής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ και που ε, προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Ήταν απολύτως σαφές ε, ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, να εφαρμοστεί η συμφωνία αυτή χωρίς ε, την σαφή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν έγκαιρα ξεκινήσαμε την διαδικασία μελέτης ε, της συμφωνίας των αξιών και των ευεργετημάτων που από αυτή τη συμφωνία μπορούν να απορρεύσουν. Ήδη σήμερα δημοσιοποίησε η Κομισιόν ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων ε, επισήμως την επόμενη εβδομάδα 17 Οκτωβρίου ε, θα επικυρώσει τη συμφωνία ε, και επομένως θα ξεκινήσει η διαδικασία επικύρωσης και στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν τούτη η ακρόαση έρχεται την κατάλληλη στιγμή πριν ακριβώς την έγκριση στο, στο Κολέγιο των ε, Επιτρόπων. Εν τω μεταξύ βέβαια την επόμενη εβδομάδα έχουμε ε, και την ε, διάσκεψη ΑΣΕΑΝ. Και επομένως αυτό... make clear that we want to have Έχουμε την άσεμ, συγγνώμη, και θα αποτελέσει ε, μια καλή, ένα καλό παράδειγμα συμφωνίας στην περιοχή ΑΣΕΑΝ. Ε, πρόκειται για ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά ε, αλλά βλέπουμε ότι κάποιοι δεν ε, σέβονται ε, πλέον αυτές τις συνολικές συμφωνίες αλλά θέλουν περισσότερο να ενδώσουν σε παιχνίδια εξουσίας. Αυτή δεν είναι η δικιά μας θέση όμως. Uh, Επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το δίκαιο και η εμπόριο Βεβαίως, πολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για τη μεταρρύθμιση του κώδικα ε, εργασίας στο Βιετνάμ, καθώς επίσης ε, και τις δεσμεύσεις όσον αφορά ε, το παράρτημα 3 της συνθήκης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, καθώς επίσης και την εφαρμογή ε, αυτή στα πλαίσια της συμφωνίας για το Κοινοβούλιο και αυτό αποτελεί βεβαίως σημαντικό θέμα. Ε, μάλιστα σήμερα το πρωί στη συζήτηση για την Ιαπωνία βεβαίως συζητήσαμε ακριβώς το γεγονός ότι η Ιαπωνία δεν έχει επικυρώσει το παράρτημα 2 της ίδιας ε, ε, συμφωνίας. Είναι σημαντικό ε, βεβαίως ότι αυτές οι συμφωνίες εμπορίου πρέπει να είναι ευεργετικές και επωφελείς για τους πολίτες και να φέρουν βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως είπα και προηγουμένως, είμαστε πεπισμένοι ότι οπωσδήποτε ε, θα είναι ιδιαίτερος ε, επωφελής ε, αυτή η συμφωνία και όχι μόνο από οικονομικής απόψεως αλλά και λόγω του ότι θα δημιουργηθεί μια καλή εταιρική σχέση. Γνωρίζω ότι πολλά ερωτήματα πέρα από το θέμα της επικύρωσης των τριών συμβάσεων του ΔΟΕ, ξέρω λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ε, τα οποία όμως θα μας συζητήσουν οι Chief Negotiators από πλευράς ε, του ε, Βιετνάμ. Έχουμε τον επικεφαλής διαπραγματευτή και επίσης έχουμε τον κύριο Τραν Κουόκ Χάν και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε την ε, κυρία Έλενα Κιόνιγκ ε, από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. καλωσορίσατε. θα έχουν και οι δύο την ε, δυνατότητα να μας δώσουν την άποψή τους σχετικά με τα ωφέλη και την αξία αυτής της συμφωνίας ε, και μετά βέβαια θα, κάνουμε και μια, ε, θα έχουμε και έναν ευρύ γύρο κατά τη διάρκεια του οποίου θα ακούσουμε εμπειρογνώμονες που θα μας δώσουν τη δικιά τους άποψη για πολλά και σημαντικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας. Να σας πω εξ αρχής ε, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι βρίσκονται εδώ και που όλοι θα έχουν την ευκαιρία και την δυνατότητα να συζητήσουν εδώ στο Κοινοβούλιο, σε αυτό το Κοινοβούλιο Ειρήνης ε, των Βρυξελών. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν όλη την δυνατότητα ε, να εκφράσουν την άποψή τους και να συμμετάσχουν στην συζήτηση. Επομένως, ε, ε, ξεκινάει επίσημα πλέον η ακρόασή μας και θα δώσω τον λόγο στον μόνιμο εισηγητή μας. Κύριε Ζαχραντήλ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω όλες και όλους Επιτροπή μας αποδείχθηκε σήμερα πόσο σημαντική είναι αλλά και πόσο σημαντικό είναι και το Βιετνάμ. Εφόσον λίγες ώρες πριν την έναρξη αυτής της ακρόασης η κυρία Μάλμστρομ, επίτροπος για τα θέματα εμπορίου, ανακοίνωσε ότι το Σώμα των Επιτρόπων την επόμενη εβδομάδα θα εγκρίνει την τελική εκδοχή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ για να ξεκινήσει η διαδικασία κύρωση. Σύμπτωση, αλλά πολύ ευτυχής. Και δίνει αυτό και σε εμά όθηση και ελπίζω να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και την ε, ευκαιρία και να ευχηθώ μια επιτυχή διαδικασία κύρωση. Ως μόνοι μουσικητές είμαι πολύ ευτυχής που άκουσα τον εαυτό και ελπίζω η όλη διαδικασία να περιγραφεί πάρα πολύ καλά εδώ στην Ακροασία. Να ότι ξεκινήσαμε με τον Ιούνιο του 2002 τις διαπραγματεύσεις. Επί της αρχής καταλήξαμε τον Αύγουστο του 2015 και τώρα μπαίνουμε τρία χρόνια μετά στην τελική φάση. Ελπίζω η διαδικασία κύρωσης να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας θητείας του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι είναι εφικτό, είναι σίγουρα ευκταίο και είναι και αναγκαίο. Γιατί, διότι αυτή η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου είναι μια σύγχρονη συμφωνία για την οικονομική ανάπτυξη. Παρέχει ένα φιλόδοξο μοντέλο εμπορικών σχέσεων και συνεργασίας με τις ανψόμενες χώρες, όπου είμαστε ισότιμοι εταίροι, έχουμε κοινούς στόχους, κοινέ αξίες, τόνωση ανάπτυξη, απασχόληση, τόνωση της ανταγωνιστικότητας, καταπολέμησης της φτώχειας και παγίωση των ε, διαθροτικών μεταρρυθμίσεων. Επιτύχαμε επίσης ε, την πιο ε, πλήρη συμφωνία ελεύθερου με μία από τις χώρες περιοχής και η οικονομική αυτή εταιρική σχέση δημιουργεί τις καλύτερες δυνατέ προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και προς οικονομικό όφελος. Ξεκάθαρα επίσης καταδεικνύεται ότι το ανοιχτό εμπόριο μαζί με τις διαρτατικές μεταρρυθμίσεις είναι ένα μέσο κοινωνικής πρόοδου, ε, ανάπτυξης ε, και σήμερα το βλέπουμε αυτό ε, γιατί η συμφωνία αυτή με το Βιετνάμ είναι μια μεγάλη επιτυχία. Πριν 30 χρόνια ήταν μια από τι φτωχότερε χώρε του κόσμου το Βιετνάμ. Σήμερα είναι μια από τι πιο δυναμικέ, ανθυρέ οικονομίε που δραστηριοποιείται στη διασυνδεδεμένη αγορά τη Ανατολική Ασία. Και η συμφωνία αυτή είναι και ένα μοντέλο για την ε, επίδειξη ήπιας δύναμης, ήπιας ισχύω. Μπορούμε να είμαστε σκαπανείς που προωθούμε το παγκόσμιο εμπόριο, το πολυμέρι σύστημα, όταν έχουμε αλλού αύξηση του προστατευτισμού, δυστυχώς. Και υπάρχουν διαφοροί ε, τομείς, λίγοι ε, που είναι πλήρως εξευρωπαϊσμένοι όπως η κοινή εμπορική πολιτική για παράδειγμα που είναι 100% ευρωπαϊκή πολιτική, λίγοι είναι οι τομείς λοιπόν που έχουν εξευρωπαϊστεί εντελώς. Μπορούμε λοιπόν να δείξουμε εδώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματική ηγεσία με στεναρό εμπόριο, με κεφάλαιο ανάπτυξης εμπορίου πολύ ισχυρό Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και κατάλληλες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Ε, έχουν αναλυφθεί δεσμεύσεις, έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα από τις αρχές του Βιετνάμ και αυτή η συμφωνία ήδη είναι ένα εργαλείο για ε, αύξηση των και αναβάθμιση των εργασιακών περιβαλλοντικών προτύπων ε, ώστε να προσεγγίσουν αυτά της Ευρώπης και το βλέπουμε από τον κώδικα ε, εργατικού δικαίου, στον τομέα της κατανοητικής παιδικής εργασίας, στον τομέα της ασφάλεια, Έχουμε θετικές εξελίξεις, υπάρχει ο δικό χάρτη, υπάρχουν δεσμεύσει και βλέπουμε ήδη και κάποια αποτελέσματα. Βέβαια, πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν. Όμως πρόκειται για μια διαδικασία διαδικασία όπου αυτή η εμπορική συμφωνία θα επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις. Δεν ε, πρόκειται για προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων. Μπαίνουμε σε μια κρίσιμη φάση, ξεκινάει περίοδος κύρωσης, όπως είπα και στην αρχή. Είναι πάρα πολύ καλή η συγκυρία. Πρέπει λοιπόν να την εκμεταλλευτούμε και να ολοκληρώσουμε το έργο μας στη διάρκεια αυτής της θητείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαραντήλ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Υφυπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου, τον κύριο Τραν Κοντακάν από το Βιετνάμ. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε της Τροπής ΙΝΤΑ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάγκε και την Επιτροπή Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσω την θέση μας, την δική μας προσέγγιση σε αυτή τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ. Κυρίε και κύριοι, όπως γνωρίζετε, το Βιετνάμ έχει προσπαθήσει να ενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία συστηματικά ακολουθώντας τους κανόνες του πολυμερού συστήματος εμπορίου και με ενεργό συμμετοχή σε πολυμερείς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς συνεργασίας. Πέραν τούτου, το Βιετνάμ είναι μέλος του ΑΣΕΑΝ, έχει επίσης συνάψει συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με πάνω από 10 εμπορικούς εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τώρα πλέον έχει φτάσει να είναι η δεύτερη πλέον ανοιχτή οικονομία στην περιοχή, με αύξηση του εμπορίου, ε, με διπλασιασμό του εμπορίου και τη συνεισφορά του στο ΑΕΠ. Το Βιετνάμ συνεχίζει να υποστηρίζει ένα ανοιχτό σύστημα διεθνούς εμπορίου βασισμένο σε κανόνες. Από το 2017 έχουμε υποστηρίξει ε, μια φιλόδοξη πολιτική εμπορικής συνεργασίας. Το Μάρτιο του 2018 το Βιετνάμ και άλλες 10 χώρες σύναψαν συμφωνία για την ε, συνεργασία στον Ειρηνικό ε, και την Νοτιοανατολική Ασία. Ε, η CPTPP, μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες που συνήφθη στην περιοχή και θα αρχίσει να ισχύει σύντομα. Θα έλεγα ότι είναι υποδειγματική για την, περίοδο, για την περιοχή μάλλον της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού σε μια περίοδο που η συνεργασία μας εμβαθύνεται κάθε μέρα. Κυρίε και κύριοι, όπως γνωρίζετε, η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Από τότε προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να ξεχωρίσει σε μια ξεχωριστή συμφωνία οι ρήτρες, οι διατάξεις για τις επενδύσεις. Αυτό το καταφέραμε τον Ιούνιο και τώρα θα, μπορέσει να θα μπορέσουν να ακολουθηθούν οι εθνικές διαδικασίες των κρατών μελών για την επικύρωση αυτών των συμφωνιών και με χαρά υποδέχομαι την είδηση ότι η Επίτροπος Μάλστρομ προωθεί την στις διαδικασίες, στην μετάφραση, όλα όσα χρειάζονται να γίνουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να επικυρωθεί η συμφωνία. Στόχος αυτής της συμφωνίας ήταν η ευάθυνση των σχέσεων. Συστηματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους του Βιετνάμ. Πάνω από 47 δισεκατομμύρια ήταν το εμπορικό μας ισογείο πέρυσι και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος των χωρών του ΑΣΕΑΝ. Και το συνεχίζεται αυτό γιατί εμπιστευόμαστε ότι και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να έχει μια μακροχρόνια σχέση μαζί μας. Πρώτος στόχος αυτών των διαπραγματεύσεων, αυτών των εμπορικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς να ενταχθεί το Βιετνάμ στην παγκόσμια οικονομία, υιοθετώντα και υλοποιώντα τους κανόνες του ΠΟΕ. Αυτό έγινε με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας στο Βιετνάμ η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικό προτιμησιακό καθεστώς. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος και το οποίο πράγματι βοήθησε έτσι ώστε το Βιετνάμ να γίνει πλέον χώρα μέσου εισοδήματο και πολλοί εκατομμύρια άνθρωποι να ξεπεράσουν το όριο της φτώχειας. Μπορούμε τώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα, πέρα από τις, το μονομερές προτιμησιακό καθεστώς και να περάσουμε σε μια αμοιβαία, ε, αποφελή ε, σχέση εμπορική και πολιτική. η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου θα εξαλείψει σχεδόν όλους τους ε, ε, δασμούς, δεδομένου ότι το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ είναι συμπληρωματικό, είναι συμπληρωματική τομή της οικονομίας που, που, στους κάθε χώρα και περιμένουμε ότι θα αυξηθεί σε απόλυτη τιμή το εμπόριο στους τομείς του εξοπλισμού, του μηχανολογικού εξοπλισμού, του τροφίμων και ποτών, ε, αγροτικών προϊόντων και άλλων. Υπάρχουν επίσης πολλοί τομείς της οικονομίας, όπως για παράδειγμα τα ποτά, ε, τα οποία μέχρι πρότινος ήταν κλειστός τομέας για ξένες επενδύσεις στο Βιετνάμ, τώρα θα ανοίξουν με τη συμφωνία. Επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα να αυξηθούν η, να αυξηθεί η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών, των ε, επαγγελματικών, των περιβαλλοντικών, της διανομής και των logistics. Επίσης, η συμφωνία περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τις δημόσιες προμήθειες με προτιμησιακό καθεστώς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το οποίο σημαίνει ότι Αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν εξαιρετικές ευκαιρίες στον τομέα των φαρακιμευτικό, στον τομέα των δημοσίων έργων και των υποδομών, των μεταφορών και άλλους τομείς. Τρίτον, χάρη στην Συμφωνία Ελευθέρου Μπορείου, οι κανόνες που έχει το Βιετνάμ όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις ε, προστατευμένων προϊόντων, την τεχνολογικά προϊόντα, την πνευματική ιδιοκτησία, αλλά και άλλους τομείς, έρχονται πλέον ε, και πληρούν τις προϋποθέσεις του διεθνούς ε, εμπορικού συστήματος. Τέλος, εξίσου σημαντικό, η Συμφορία Ελευθέρων Εμπορίου καλύπτει ευρύτατες τομείς και σημαντικές δεσμεύσεις και για τους δύο εταίρους στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος. Το οποίο σημαίνει ότι η αύξηση αυτού του εμπορίου και η ανάπτυξη που περιμένουμε θα γίνει ταυτόχρονα με την προσπάθειά μας για φορεία. Ελπίζουμε ότι αυτή η σχέση, η κοινή σχέση των Βιετναμέζων και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Είναι πολύ θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σύναψε τέτοια συμφωνία που κοιτάει προς το μέλλον με μια αναπτυσσόμενη χώρα στην περιοχή αυτό ανοίγει μεγαλύτερε προοπτικέ για τι εμπορικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε τη περιοχή. Κυρίε και κύριοι, η σύναψη εμπορικών συμφωνιών είναι σημαντική από μόνη τη, αλλά είναι απλώ το πρώτο βήμα. Η κυβέρνησή μου έχει ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζεται για το σχέδιο εφαρμογή τη συμφωνία, η οποία θα υποβληθεί στο Εθνικό μα ε, Κοινοβούλιο, έτσι ώστε και οι επιχειρήσει και οι πολίτε και των δύο μερών τη συμφωνία να υποφεληθούν από αυτή. Ειλικρινά ελπίζω ότι σε λίγα χρόνια η επόμενη γενιά θα μας ευγνωμονεί για αυτές τις αποφάσεις, για αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζουμε προς όφελος των πολιτών μας και στέλνοντας ένα ξεχάθαρο μήνυμα στο διεθνή σκηνικό, στο διεθνές επίπεδο, εναντίον του προστατευτισμού. Είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε στην παγκόσμια οικονομία ως ανοιχτό κράτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καν. Και τώρα από την ε, ευρωπαϊκή πλευρά η Έλληνα Κρούγκερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Πρόεδρε Λάγκερ, κύριε Ισαγητά, μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Χάν για να συζητήσουμε αυτήν την Συμφωνία Εμπορίου και ε, ε Επενδύσεων. Δύο συμφωνίες που συζητήθηκαν ε, μαζί. Όντως, ε, η απόφαση να παρουσιαστούν τα δύο θέματα μαζί ήταν πολύ σωστή πολύ κατάλληλος ο χρόνος ε, διεξαγωγής αυτής ε, της ε, ακρόασης. Θα ήθελα να ασχοληθώ με την συμφωνία, κυρίως πρώτα όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία για τους εξαγωγείς και τους επενδυτές. Όταν άρχισε να βγαίνει η χώρα από μια μακρά περίοδο ένδυας και αποκλεισμού, ε, διαπιστώσαμε ότι η χώρα έχει ξεκινήσει να αλλάζει κοινωνικά και οικονομικά ε, ε, και παράλληλα με την πορεία ένταξης, όπως είπε και ο Υπουργός προηγουμένως, της χώρας στην οικονομία την παγκόσμια οικονομία. Μιλάμε τώρα για 95 εκατομμύρια ε, ανθρώπους ε, με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Ε, επίσης μιλάμε για μια χώρα η οποία μέχρι ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει εκριζώσει την μεγάλη φτώχεια σε σχέση με την ε, περιοχή Ασιάνα ε, το Βιετνάμ έχει καλή συνδεσιμότητα με άλλες μεγάλες χώρες της περιοχής. Είναι μία από τις ε, ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες της περιοχής με ρυθμό ανάπτυξης 6% τις τελευταίες δεκαετίες. Η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη του Βιετνάμ έχει οδηγήσει και σε ε, ε, καλές ε, συμφωνίες και εμπορικές σχέσεις. Η συμφωνία η οποία άρχισε να υλοποιείται το 2016 ήταν ένα ισχυρό πρώτο βήμα. Όπως υπόθηκε, το Βιετνάμ είναι ο δεύτερος μεγάλος μας εταίρος ε, ε, στην Ασία μετά τη Σιγκαπούρη και πριν από την Μαλαισία. Βεβαίως 8,2 8,3 δις ε, είναι το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών, ωστόσο αυξάνονται διαρκώς ε, και οπωσδήποτε θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πλατφόρμα επί της οποίας θα βασιστούμε για να αναπτύξουμε περαιτέρω ε, τις σχέσεις. Όσον αφορά τώρα τη στρατηγική σημασία αυτής της συμφωνίας, γιατί θα πρέπει να την εντάξουμε στο ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά τρίτες ε, χώρες με τις οποίες ε, το Βιετνάμ ε, έχει συμφωνίες είναι το ΑΣΕΑΝ, Κίνα, Ινδία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κορέα και η Ιαπωνία με τις οποίες έχουν διμερείς με την ομάδα ΑΣΕΑΝ και αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε την εταιρική σχέση καθώς επίσης και την CTPPT ή την ενδεκάτη στη σειρά ε, συμφωνία. Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ε, θα δώσει την δυνατότητα να επιρρευθεί το επίπεδο των ε, ανταγωνιστών μας στην περιοχή και ε, σε ορισμένες περιπτώσεις ε, να το ε, ξεπεράσουμε. Η συμφωνία με την Κορέα, την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη, λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλάμε για την Νοτιοανατολική Ασία και μετά κυρίως από τη συμφωνία με την Σιγκαπούρη, ετέθη ο ακρογωνιαίος λήθος για τις σχέσεις με την περιφέρεια αυτή, έτσι ώστε ε, να φτάσουμε κάποια στιγμή σε region to region συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΑΣΕΑΝ. Ε, βεβαίως το Βιετνάμ αποτελεί ε, και η συμφωνία με το Βιετνάμ λόγω ακριβώς ε, του φιλόδοξου σχεδιασμού του μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες συμφωνίες με την Μαλαισία ας πούμε. Όπως αναφέρθηκε άλλωστε και σε προηγούμενες παρεμβάσεις θέλουμε εδώ να δώσουμε κάποιες γενικότερες κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να κάνουμε ε, και να ασκήσουμε το διεθνές εμπόριο, αντίθετα από τα όσα αυτή την περίοδο συμβαίνουν. Επί της ε, ουσίας και μάλιστα ο Υπουργός ο ε, κύριος Χάνε αναφέρθηκε σε πολλά από τα θέματα αυτά. Πρόκειται για την πιο πλήρη και φιλόδοξη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την ε, φιλοδοξία που είχαμε με την ε, Σιγκαπούρη. Κυρίως όμως ε, πρόκειται για μια συμφωνία την οποία εμείς έχουμε σχεδιάσει ως δυνάμενη να εξελιχθεί, ακολουθώντας δηλαδή και τις λοιπές εξελίξεις αναφέρθηκε ότι σε 7 χρόνια θα έρθουν οι τα δεσμολογικά εμπόδια Ε, πολλά, πολλοί, από τους εξαγωγικούς, ε, πολλοί από τους δασμούς επίσης ε, θα σταματήσουν να ισχύουν. Θα ωφεληθούν μικροί γεωργοί και μικρές εκμεταλλεύσεις κυρίως στα πλαίσια της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, θα υπο, ε, θα, θα προωθηθούν στοιχεία τα οποία αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη καθώς επίσης και το, την οικολογική αντιμετώπιση. Αυτό το FTA, δηλαδή Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, ε, θα ε, αφορά και υψηλής ποιότητας επενδύσεις που είναι ευχή και των δύο πλευρών. Έρχομαι λοιπόν στο IPA. Ε, πρόκειται το EPA ε, το οποίο ε, πρόκειται, είναι μια συμφωνία η οποία πρόκειται να υπογραφεί και η οποία δίνει υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδύσεων, κυρίως θέτοντας συγκεκριμένα υψηλά πρότυπα η νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστασία ε, των επενδύσεων προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα ε, στην προστασία των θέσεων εργασίας και την ποιοτική εργασία αφενός και την ε, αρμοδιότητα και δικαιοδέσια που έχουν η κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις. Επίσης το θέμα επίλυση των διαφορών είναι ένα σημαντικό σημείο. Υπάρχει δεσμευτικός κώδικας συμπεριφοράς ε, για τα μέλη, καθώς επίσης ε, και ε, κανόνες μεσολάβησης. Όσον αφορά τις αξίες τώρα, γιατί συζητούμε για ωφέλη και αξίες η πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ε, λέει ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξει μαζί με τις εμπορικές συμφωνίες και προστασία του περιβάλλοντος ε, και της εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε βιώσιμη ε, ανάπτυξη με υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Ε, δεσμεύσεις και καθήκοντα λοιπόν για προστασία των θεμελιδών ε, δικαιωμάτων ε, και των κανόνων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι ανεξάρτητοι ε, εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί έτσι ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο της ε, συμφωνίας με το ε, Βιετνάμ και σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτό ήταν μία από τις εστιάσεις μας. Μία στρογγυλή τράπεζα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την βιώσιμη ανάπτυξη έλαβε χώρα το Μάιο του 2000, τον Μάιο του 2015 ε, και εκεί συζητήθηκαν ε, και τα στοιχεία ε, της συμφωνίας που αφορούν ακριβώς τα θέματα αυτά και ο τρόπος αντιμετώπισης ε, των ε, ζητημάτων αυτών που θεωρούνται πολύ σοβαρά ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι βεβαία ότι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου θα οδηγήσει σε βελτίωση όλων των θεμάτων αυτών και σε επικύρωση των συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και ταυτοχρόνως προβλέπεται και δέσμευση και εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. και μέσω του PCA, του FTA και των εξειδικευμένων ε, επιτροπών θα υπάρξει προώθηση ε, της ε, συμφωνίας και με τον τρόπο αυτό έρχομαι και στα επόμενα βήματα. Προχωράνε οι διαπραγματεύσεις για την συμφωνία και όπως είπε και ο Υπουργός κύριος Χάν προχωρούν ε, και ε, οι επιμέρους, τα διαδικαστικά της συμφωνίας. Μεταφράζεται η συμφωνία σε όλες τις γλώσσες. Και πολύ σύντομα θα δοθούν στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Επίσης προσπαθούμε να αξιολογήσουμε ε, τα, ε, όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όταν θα επικυρωθεί η συμφωνία θα ξέρουμε ξεκάθαρα ε, τι χρειάζεται να κάνουμε και τι έχουμε ήδη υλοποιήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα καταρχάς το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κύριο Παντζέρη, για δύο λεπτά και εν συνεχεία στον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας ε, με την Νοτιοανατολική Ασία για δύο λεπτά. Και μετά θα ε, δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. 15 λεπτά έχουμε για αυτή την ε, συνεδρία ερωταπαντήσεων. Κύριε Παντσέρη. Α, θέλετε να δώσω το λόγο στην κυρία Λοχμπίλερ. Εντάξει, ακούσουμε την κυρία Λοχμπίλερ. Ναι, συνεργαζόμαστε, λέει η κυρία Λοχμπίλερ. Οπότε θα περάσω εγώ το μήνυμα. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ε, σε σχέση με τις ε, δεσμεύσει που είχαν λάβει η χώρα να σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι πολύ αυστηρές ε, οι διατάξεις ε, για τα ασφαλεία. ασφαλείας. Γι' αυτό υπάρχουν καταστολέ, έχουμε διώξει ανθρωπίνων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ της έχει ζητηθεί να μην ε, διώκει τις οργανώσεις κοινωνικών πολιτών και του υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εμπειρογνώμονε, οι οποίοι εξέφρασαν ε, ανησυχίε για το πώς αντιμετωπίζονται οι ειρηνικοί διαδηλωτέ. Υπήρχε το άρθρο 79 ε, του ποινικού κώδικα του 1999, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να τους καταδικάσει τους αντιφρονούντες και τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει δε το άρθρο 79 ε, αναφορά και σε πιθανή καταδίκη στα θανατική ποινή. Ο κύριος ε, Πουεντσέρη εκφράζει την μεγάλη ανησυχία σε σχέση με αυτή τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών, ε, ακριβώς λόγω του προβλήματος με το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε μείζονε τομεί εξαγωγή επίση, όπω είναι ο τομέα εισφασμάτων κλεισοφαντουργία. Επίση, εδώ έχουμε προβλήματα. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητα συνδικάτα. Το δικαίωμα στην απεργία είναι περιορισμένο και απαγορεύεται μάλιστα ε, κάθετα σε διάφορε τομεί. Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου περιλαμβάνει αδυναμίε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα σε σχέση με την ε, Trans-Pacific Partnership ε, για χώρες που περιλαμβάνουν και τη ΣΥΠΑ μεταξύ άλλων και χώρες του ειρηνικού Ξέρουμε ότι με την τελευταία αυτή συμφωνία ε, CTPP υπάρχουν θετικά στοιχεία. Έχουν αναλυφθεί υποχρεώσει για βελτίωση τη κατάσταση των αρέσεων δικαιωμάτων. Έχουμε την 87, ε, 97 και 105 συμβάσει του ε, Διεθνού Οργάνωση Εργασία που υποτίθεται ότι θα τεθούν σε ισχύ πριν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Θα κυρωθούν δηλαδή τρει αυτέ. Αλλά δεν προβλέπεται αυτό στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με το Βιετνάμ. Και η ερώτηση είναι και προς τον Υφυπουργό. Οι τρεις συμβάσεις του ΔΣΔΟΕ θα γίνουν εθνικό δίκαιο πριν ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη συμφωνία αυτή ελεύθερων συναλλαγών. Και έρχομαι στην κυρία Κένιχ να κάνω το εξή ερώτημα. Εσώσουμε σε ανθρώπινα δικαιώματα και η σύμβαση της ΔΟΕ. Γιατί δεν μπήκε ως προαπαιτούμενο πριν τη σύναψη της ε, ολοκλήρωσης αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ κύριος ε, Λάγκεν. Εσείς έχετε τώρα το λόγο που είστε πρόεδρος Επιτροπής με, για τη σχέση με την Ανατολική Ασία. Ναι, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να τοποθετηθώ και εγώ ως πρόεδρος ε, της Αντιπροσωπείας για τη σχέση με τις χώρες ε, και είμαι ευρωβουλευτής. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη η πρόοδος που θέλουμε να επιτύχουμε μέσω αυτής της συμφωνίας. Υπήρξαν διάφορες συζητήσεις, είχαμε τη Σιγκαπούρη, ε, ολοκληρώθηκαν και διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α, Έλεγα λοιπόν ότι για μας είναι σημαντικό όταν αλλάζει άρδιν ε, η παγκόσμια εμπορική πολιτική, όταν έχουμε αυτές τις ε, ε, θέσεις, σχέσεις, τις διμερείς με τις χώρες σας που θέλουμε να ενισχύσουμε, έχει μεγάλη σημασία αυτή η συμφωνία που θέλουμε να είναι ένα σημείο αναφοράς για τις χώρες περιοχής και με τη Φιλιππίνες, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, την θέλουμε σε ένα άλλο στάδιο να προχωρήσουμε σε αντίστοιχες συμφωνίες και έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη είναι η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη στο Βιετνάμ. Έχουμε ένα νέο πληθυσμό σε ηλικία ε, σταθερό, έχουμε εργαζόμενους, ε, εργατικούς εργαζόμενους θα έλεγα ε, και καλό είναι να βαθυνθούν οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να δούμε όμως τι γίνεται με το πολιτικό σύστημα Σίγουρα δεν θέλουμε να μπούμε στα ιδιωτικά και στα εσωτερικά ε, δεν είναι το μονοκομματικό σύστημα του Βιετνάμ κάτι που εμείς το ε, έχουμε ως σύστημα δικό μας εδώ, αλλά αυτό που είπε και η κυρία Λοχμπίλερ, ε, θέλουμε τη Συμφωνία Ελεύθερων αλλαγών θέλουμε να την υποστηρίξουμε, όμως γι' αυτό υπάρχουν προαπαιτούμενα κατά εμάς. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα εργασιακές συνθήκες, τι γίνεται με τους προσφέρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θέλω και εγώ να τονίσω το εξής ερώτημα. Πώς τα βλέπουμε Βλέπετε πριν εμείς περάσουμε ε, ως κοινοβούλιο στην κύρωση αυτή ε, την ε, ε, συμφωνία, πώς θα την εντάξετε στο Εθνικό Δίκαιο και ιδίως τι θα γίνει με το διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. πρέπει να γίνει απτή πρόοδος και σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφραση, ελευθεροτυπία, τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, και πραγματικά παρά την εφορία από τα καλά νέα, ε, ε, αυτά τα θεωρώ απολύτω απαραίτητα. Και την κυρία Κένιξ, ό,τι αφορά τη βάση των δύο συμφωνών που διαπραγματεύω, μήπως θα μπορούσε να γίνει μια γενικότερη συμφωνία. for the floor. Reach to reach. Ε, τώρα έχω, βλέπω, 6-7 συναδέλφους που ζητούν το λόγο. Λοιπόν, 1,5 λεπτό ο καθένας. Πρώτη Μαρία Ρενά. Ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι κι εγώ μεταξύ των 32 ευρωβουλευτών που έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις ανησυχίες μας για αυτήν τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ ανησυχίες οι οποίες σχετίζονται ιδιαίτερα με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ, με την ελευθερία της εκφράσης, με τη λογοκρισία, με την μη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, με τις διώξεις συνδικαλιστών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το άρθρο 3 της Συμφωνίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιβάλλει να προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα με όλες τις πολιτικές μας. Και θέτω το ερώτημα λοιπόν στην Επιτροπή. Θεωρείτε ότι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, την οποία έχετε διαπραγματευτεί με το Βιετνάμ, είναι συμβατή με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο ερώτημα και πάλι στην Επιτροπή. Μιλήσατε για τις επενδύσεις, το κεφάλαιο για τις επενδύσεις, η οποία ε, προβλέπει και πάλι ένα ICS, ένα δικαιωτοδοτικό όργανο. Το οποίο σημαίνει ότι αν κάποιος επενδυτής στο Βιετνάμ θεωρεί ότι ευλάφθηκε, μπορεί να προσφύγει σε ένα ιδιωτικό, διαφορετικό, παράλληλο δικαιωτικό όργανο. Θέλω να μου πείτε το εξή. Μετά τους διώξεις και τους φυλακίσεις συνδικαλιστών, υπάρχουν βεβαίως διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αφαιρθεί το Βιετνάμ μπροστά στους επενδυτές και εκείνοι θα έχουν ένα δικαίωμα προσφυγής εναντίον της απόφασης ή της πολιτικής του Βιετνάμ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια αντίστοιχη δυνατότητα προστασίας των συνδικαλιστών. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Η κυρία Καρτον η ερώτηση και η δική μου είναι παρόμοια και εγώ είμαι ανάμεσα στους 32 ευρωβουλευτέ που έστειλαν αυτή την επιστολή. Ήμασταν από όλα τα πολιτικά κόμματα, από όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου. Πριν την προσχώρηση του Βιετνάμ στον ΠΟΕ, είχε αναλάβει ορισμένε δεσμεύσει σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα ήδη από τότε. Όμω οι πληροφορίε που έχουμε για την κατάσταση στο Βιετνάμ από τι οργανώσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του υπερασπιστέ του είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, ότι υπάρχει περισσότερη καταστολή ε, με το νομοθεσία, για παράδειγμα, για το διαδίκτυο, με ε, επιβολή ποινών σε υπεράσπιτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με άλλου τύπους διώξεις, όπως για παράδειγμα να μετατίθενται άνθρωποι, ε, να μεταγάγονται μάλλον άνθρωποι σε φυλακές μακριά από τις οικογένειές τους, έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο ε, δύσκολη η ποινή τους. Θέτω λοιπόν αυτά τα ερωτήματα και το ερώτημά μου είναι τι ζητάει, τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβεί πριν να φτάσουμε σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι περιμένει να γίνει η Κομισιόν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και προς τις αρχές του Βιετνάμ. Ποιος είναι ο δικός σας χάρτης. Άκουσα πολλές φορές να, αναφέρεις, να αναφερόμαστε στην βιώσιμη ανάπτυξη και στα, και στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Όμως, για εμένα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα είναι εξίσου σημαντικά με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα χωρί να υπάρχει πραγματική ελευθερία τη έκφραση. Δεν μπορεί κανεί λοιπόν να ε, σπάει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ορισ... και να προσπίζεται μόνο ορισμένα. Θα πρέπει λοιπόν να αναλυφθούν ουσιαστικέ δράσει κατά την άποψή μου άμεσα, το οποίο σημαίνει απελευθέρωση κρατουμένων συνείδησης, πολιτικών κρατουμένων, να απελευθερωθεί η δυνατότητα κάποιων να δημοσιοποιούν τη θέση τους online, οι bloggers, έτσι ώστε τα λόγια να γίνουν πράξη. Γιατί διαφορετικά θα, δεν θα ήθελα να επαναληφθεί αυτό που συνέβη πριν την προσχώρηση στον ΠΟΕ του Βιετνάμ, το οποίο ανέλαβε πολλές δεσμεύσεις στα λόγια, αλλά τίποτε δεν άλλαξε στην πράξη. Ναι, ακούσαμε πολλά κυρία Κασβάντερ. Το εμπόριο είναι σημαντικό και σίγουρα το ε, ε, ενστερνιζόμαστε κι εμείς. Αυτή η εμπορική συμφωνία θα είναι ένα νέο μοντέλο εμπορικής πολιτικής Υπάρχουν ε, επικεφαλίδες και τίτλοι, αλλά μου λείπει το περιεχόμενο. Ακούσαμε διάφορα, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, για παράδειγμα, ή τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εκεί βλέπουμε ανάγκη να γίνουν πολλά ακόμη. Επίσης, ε, ε, ο κύριος Λάγκεν ανέφερε και για άλλες ε, περιπτώσεις. Ε, έχουμε και την Ιαπωνία, έχουμε και το Βιετνάμ και άλλη μια περίπτωση. Ε, πρέπει να μου πείτε επίσης αν η χώρα σας θα κυρώσει τις τρεις συμβάσεις της ΔΟΕ. Επίσης, το κεφάλαιο της βιωσιμότητας. Δεν υπάρχει μηχανισμός επιβολής κυρώσεων. Τι θα γίνει αν υπάρξει κάποια παράβαση. Και μια γενική ερώτηση συγκεκριμένα. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι είστε διτεθειμένοι να κάνετε για να δείξετε ότι είστε προσιλωμένοι προς το στόχο αυτό. Και ότι λαμβάνετε υπόψη σοβαρά αυτά που εμείς εκφράζουμε ως ανησυχία. Χάιντι Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ε, ασχοληθώ με την ιδιαίτερη ε, φύση ε, το Voluntary Partnership Agreement με το Βιετνάμ που μας έχει απασχολήσει στην Επιτροπή μας και είμαι μάλιστα η συγγήτρια. Ε, μου είναι ιδιαίτερος προσφυλές το εργαλείο αυτό γιατί έχει αποδείξει ε, ότι είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους ενθάρρυνσης ε, των νόμιμων εξαγωγών ξυλίας και νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος μέσω του οποίου το Βιετνάμ μπορεί να ε, ε, διασφαλίσει ότι νομίμως εξάγονται ε, τα προϊόντα γελοτομίας. Πρέπει όμως να είμαστε βέβαιοι ότι ε, και στο Βιετνάμ ε, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες νομοθετικές ε, μεταρρυθμίσεις και ρυθμίσεις για την διασφάλιση ακριβώς της νομιμότητας των προϊόντων υλοτομίας και ξυλίας. Γιατί διαφορετικά ενδεχομένως θα έχουμε τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που θα κορυφώσει τις ε, προσπάθειές μας, ε, ε, αλλά δεν θα, δεν θα είναι πλήρης εάν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά την ξυλία. Και μια σημαντική ερώτηση για την Κομισιόν, γιατί εγώ είμαι η συγκήτρια για το Voluntary Partnership Agreement. Η εισαγωγική δασμή για αυτά τα προϊόντα ξυλίας θα απελευθερωθούν πλήρως όταν η Συμφωνία Ελευθερών Εμπορίου θα τεθεί σε ισχύ. Ερωτηματικό. Ναι, συνεχίστε παρακαλώ κύριε Χαουτάλα. Είναι πιθανό να χάσουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε το θέμα των, της νομίμως ε, υλοτομηθής της ξυλίας. Πρόεδρος. Παρακαλώ πολύ να μην ξεπερνάτε το χρόνο μιλίας. Αναφυσβήτητα όλοι έχουν πολύ σημαντικά θέματα να ρωτήσουν. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθεια έτσι ώστε να έρθουν εδώ. Επομένω, ο κατάλογο αγορητών ε, ε, έχει κανονιστεί. Παρακαλώ να μην ξεπερνάτε το χρόνο Αλέσια Μόσκα. Είναι προφανέ από τους προναλύσαντε ε, ότι το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα. Αυτό με κανένα τρόπο δεν, θε, δεν ε, έρχεται για να μειώσει την αναγνώριση της σημασίας αυτής της ε, συμφωνίας και αναγνωρίζουμε τη γεωπολιτική στρατηγική ε, σημασία της συμφωνίας. Ωστόσο, η Βιετναμέζικη κυβέρνηση οπωσδήποτε θα πρέπει να δώσει ε, ε, σημεία και μηνύματα ότι ε, έχει ανακρούσει πριν όσον αφορά ορισμένα θέματα. θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα και τα πολιτικά δικαιώματα. Αλλά αντί να γίνονται βήματα προς τα εμπρός, βλέπουμε όπου στοχώρηση για τα θέματα αυτά είναι σημαντικό να δείξετε ότι έχετε την ικανότητα και έχετε την βούληση να εμπλακείτε με πιο συγκεκριμένο τρόπο και μέσω συγκεκριμένων δράσεων, ε, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναγνωριστεί. Και μάλιστα μιλάμε για δράσεις οι οποίες δεν απαιτούν μεγάλη ε, νομοθετική μεταρρύθμιση, ας πούμε απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων ή τροποποίηση ε, της νομοθεσίας για την κυβερνοασφάλεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Φεράντσα. Ε, ε, ορισμένοι από τους, ε, λέει η κυρία Φορέντσα, από τους προλαλήσαντες η κυρία ε, Αρένα, ας πούμε, είπαν αυτά που ήθελα και εγώ να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την δυνατότητα που μας ε, δίνεται για ανταλλαγή απόψεων με το Βιετνάμ, που είναι μια χώρα που τις τελευταίες δεκαετίες είδε πολύ μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης που οδήγησε εκτός της φτώχειας πάρα πολλούς ανθρώπους. Την προηγούμενο Ιουνίου ξεκίνησαν διαμαρτυρίες ε, του πληθυσμού για την, κατά της δημιουργίας ε, ε, ζωνών οικονομικού ενδιαφέροντος Υπάρχουν ήδη 18 οικονομικές ζώνες ε, στην χώρα και λαμβάνοντας υπόψη ότι ε, ήδη αυτές ε, προσελκύουν ξένους επενδυτές. Θεωρείτε ότι επιπλέον ζώνες θα διατηρήσουν ένα καλό επίπεδο όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Επίσης, εμείς ζητούμε από το Βιετνάμ ε, να ε, επικυρώσει και να υπογράψει όλες αυτές ε, τις συνθήκες του ΔΟΕ, κυρίως δε αυτήν με τη, για την ελευθερία του συνεταιρίζεστε και της εργασιακής εκπροσώπησης. Επίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει συγκεκριμένα μέτρα η κυβέρνηση του Βιετνάμ έτσι ώστε να συμμορφωθεί με τις συμφωνίες των Παρισίων. Και επίσης να, να γίνουν σεβαστά και τα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φιέλνερ, ορισμένοι από τους σοσιαλιστές ιδιαίτερα συνάδελφους έκαναν σχο... Ε, αναφορές στη TPP. TP. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ το κεφάλαιο το σχετικό με τις προϋποθέσεις είναι ευρύτερο, ιδίως όσον αφορά το περιβάλλον. Μετά έχει τεθεί το ζήτημα των κυρώσεων. Θέλω να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν έχουμε οποιαδήποτε, υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία εμπορίου οπουδήποτε στον κόσμο που να έχουν προβλεφθεί τέτοιες κυρώσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Και τρίτο ερώτημα, το οποίο είναι ευρύτερο, θα ήθελα να ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να πούμε ότι είμαστε λιγότερο γενναιόδοροι, τουλάχιστον όσον αφορά την κλωστή φαντουργία και τα, τα, τα ρούχα, όταν πλέον τους δίνουμε τη δυνατότητα να πάνε πέρα-πέρα, να χρησιμοποιούν πηγές πρώτων από περισσότερες από μια χώρα, από ότι, κάτι που δεν προβλεπόταν στο γενικό προτιμησιακό καθεστώς. Γιατί λέμε ότι αυτό είναι πιο αυστηρό, λοιπόν. Τέλος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει σεβασμός του κράτη δικαίου σε αυτή τη χώρα. Επομένως, είναι ουσιαστικής ε, σημασίας το ζήτημα της δικαιοδοσίας. Όμως είναι λογικό να περιμένουμε ότι ένας επενδυτής θα επιλέξει εκείνον που θα επιλύσει τη διαφορά του ε, όχι ελεύθερα, αλλά από έναν κατάλογο που θα έχει καταπτύσει το Βιετνάμ. Ευχαριστώ. Κύριος Λάγκε, σας ευχαριστώ. Θα δώσω του λόγο στους ε, διαπραγματευτές μας, μάλλον με την αντίστροφη σειρά, ξεκινώντα από την κυρία Κιόνιχ. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να είστε σύντομοι. Κύριε Κιάννη, θα προσπαθήσω. Για να... Αυτό μου σημαίνει ότι σημαίνει κάποια θέματα για να απαντήσει ο Υφυπουργό Χάν, Χάν, αλλά εν πάση περιπτώσει ετέθησαν πολλά ζητήματα και προ τον ίδιο. Ξεκινώ με το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίω, συμφωνούμε όλοι ότι η κατάσταση δεν είναι ιδανική με ελάχιστε από τι χώρε με τι οποίε έχουμε εταιρική σχέση, ακόμα και με τα κράτη-μέλη μα δεν θα μπορούμε να πούμε ότι είναι τα πράγματα ιδανικά. Βέβαια, πρέπει να λάβει κανεί υπόψη του από πού ξεκινούμε και πού πηγαίνουμε. Δηλαδή, ποια είναι η τάση. Και εμεί το βλέπουμε διαφορετικά. Πώ μπορούμε να ενθαρρύνουμε μια θετική τάση, με τάση βελτίωση τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεδομένου μάλιστα ότι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου καλύπτει και άλλα ζητήματα όπω το περιβάλλον και τα εργατικά δικαιώματα, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν το κοιτούμε ξεχωριστά. Στην συμφωνία ε, ε, για τις επενδύσεις που έχει ήδη τελειώσει η πραγματευτή της είχαμε ουσιαστικό κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν σχετικές αναφορές και στη συμφωνία για το εμπόριο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες από τους συναδέλφους, τους προσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Χανόη, έτσι ώστε να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι που είναι μια γενικότερη, ευρύτερη πολιτική της Ένωσης. Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα μάλλον, το μηνύματα που έχουμε από το Βιετνάμ είναι ότι θα επιδιώξει την επικύρωση των τριών συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Ελπίζω, φαντάζομαι, ότι θα επανέλθει και από αυτού ο Υφυπουργό της Κυβέρνησης του Βιετνάμ το παρακολουθούμε το θέμα, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος προς την επικύρωση αυτών των συμβάσεων. Γενικά μιλώντας λοιπόν, στόχος μας είναι να δούμε αυτά αποτελέσματα βέβαια, αλλά το θέμα είναι να δούμε την μεταβολή, την τάση, Σίγουρα δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Το θέμα, αυτό και αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι κάτι θετικό όσον αφορά τις συμβάσεις του ΔΟΕ. RTSD. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ευρύτερο από το αντίστοιχο κεφάλαιο της CPTTP. Δεν θα ήθελα να ξανανοίξουμε την συζήτηση για τις κυρώσεις. Θα είδατε εξάλλου και το σχέδιο δράσης με τα 15 σημεία, το οποίο ήδη προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε, κάνοντας μια παρακολούθηση του εάν θα ε, ε, ε, εγκριθούν αυτές τις συμβάσεις του ΔΟΕ, παρακολουθώντας τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Κοιτούμε δηλαδή όλα τα ζητήματα που καλύπτονται στο κεφάλαιο TSD και χαίρομαι επίσης που σε αυτή την εμπροϊκή συμφωνία προβλέπεται ρητά και δέσμευση του Βιετνάμ και των δύο μερών να ε, εφαρμόσουν τη Συμφωνία των Παρισίων. Τώρα, όσον αφορά τα βασικά ζητήματα, το, την καταπολέμηση της παράνομης πράγματι, όταν ε, τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία θα απελευθερωθεί αυτό το εμπόριο. Όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης έχει σχετική δέσμευση το Βιετνάμ συζητιέται το ενδεχόμενο να υπογράψει την Διεθνή Σύμβαση. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι, και θα το πω ειλικρινά, δεν θα χάσουμε τη δυνατότητά μας να ασκήσουμε πίεση προς αυτή την κατεύθυνση με την απελευθέρωση του εμπορίου. Το Βιετνάμ έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να προσυπογράψει τις συμβάσεις FLECT για την καταπολέμηση της παράμονης ε, ε, υλοτομίας έχει και το ίδιο, είναι και προς το συμφέρον του ιδίου να προστατεύσει το περιβάλλον και τα δάση του. Θα έλεγα ότι όσο πιο γρήγορα συμβεί αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε και το πρόβλημα και την καταπολέμηση του προβλήματος της παράνομης ε, υλοτομίας. Και κλείνω με το ερώτημα που μετέθη εάν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ κυρώσει που προβλέπονται σε κεφάλαιο TSD γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει προσφυγές με βάση άλλα κεφάλαια. Ποιο είναι το θέμα. Δεν έχει υπάρξει καμία προσφυγή στην οποία ο να μπορέσει να αποδείξει ότι υπάρχει ουσιαστική σχέση μεταξύ της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από το κεφάλαιο TSD που να είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στην επένδυσή του ή στο εμπόριο. Γι' αυτό λοιπόν δεν ευδοκίμησε καμία από αυτές τις προσφυγέ και άρα δεν είχαμε κυρώσει. Πιστεύουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε είναι η συνεργασία και γι' αυτό προτείνουμε ένα σύστημα στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εφαρμογή της συμφωνίας ένα σύστημα συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο, γιατί εκεί γίνεται μια συζήτηση μεταξύ των κυβερνήσεων, με συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών, με συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμών και με δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Γνωρίζω ότι υπάρχουν διστάμενε απόψεις για το θέμα αυτό, αλλά τουλάχιστον αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι το αποτέλεσμα των πραγματεύσεων ήταν αυτό που ήταν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα σας τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας, αγαπητοί βουλευτές. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να είμαι σύντομο, εφόσον είναι τόσο πολλά αυτά τα ερωτήματα που απευθύνθηκαν σε μένα. Θα κάνω ό,τι μπορώ Πάντως, για να σας τα εξηγήσω όλα. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά ζητήματα, για μα είναι η πρώτη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που περιλαμβάνει ισχυρή δέσμευση για το σεβασμό, την προώθηση και την αποτελεσματική εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των εργοσιακών όπω ε, ε, τα κατοχυρώνει η σύμβαση της ΔΟΕ και έχουμε πει ότι κάθε πλευρά θα κάνει συνεχείς προσπάθειες προς την κύρωση, εφόσον δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, ε, των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ. Από τότε που έγινε αυτή η δήλωση και τις δύο πλευρές, εμείς ε, υπεγράψαμε μία πλήρη συμφωνία, το Trans-Pacific Agreement, με παρόμοιες δεσμεύσεις και θέλω να σας επιβεβαιώσω ότι στην CTPPP δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να απαιτεί νομοθετικές αλλαγές πριν την έναρξη ισχύω αυτής της συμφωνίας CPTPP. Στη δική μας την περίπτωση και ακόμη και παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπογραφεί ακόμη η Συμφωνία Ελευθερομπορίου με την Ένωση, Προετοιμαζόμαστε ενεργά ήδη από τώρα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει ε, στο πλαίσιο του χάρτη βιώσιμης ανάπτυξης αυτής της συμφωνία και μπορώ να σας το πω ήδη αυτό. Μετά την σύναψη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργό του Βιετνάμ ενέκρινε το Δεκέμβριο του 2015 ήδη ε, με διάταμα ένα με νόμο τέλος πάντων την ε, ε, επικύρωση των τριών συμβάσεων που δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί από την Εθνοσυνέλευση του Βιετνάμ. Από τις οκτώ συμβάσεις της ΔΟΕ, πέντε τις έχουμε ήδη κυρώσει, τρεις παραμένουν, έχουμε το χρονοδιάγραμμα για να προχωρήσουμε στην κύρωση και αυτών και περιλαμβάνει συγκεκριμένες προσπάθειες από πλευρά της ε, κυβέρνησης σε αυτό το διάγραμμα και για τη διάδοση πληροφοριών. Την ένταξη των διεθνών αρχών στο βιετναμέζικο δίκαιο, δημιουργία υποδομών, ικανοτήτων για την κυβέρνηση κτλ. Επίσης υπάρχει πρόταση της κυβέρνησης προς ε, την Εθνοσυνέλευση για αναθεώρηση του εργατικού κώδικα, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της ΔΟΕ. Και αναμένεται ότι θα υποβληθεί αυτός ο αναφερμένος νόμος το Μάιο στην Εθνοσυνέλευση και θα τεθεί σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2019. Η κυβέρνηση τώρα, με τη βοήθεια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και άλλους ε, δωρητές ε, σύμφωνα με το νομοθετικό πρόγραμμα, όπως αυτό το αποφάσισε η Εθνοσυνέλευση, προχωρά τις σχετικές εργασίες και θέλω να σας πω ότι παρότι δεν έχει ακόμη υπογραφεί η Συμφωνία Ελεύθερου ήδη γίνονται βήματα στο Βιετνάμ για να είναι σεβαστές οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο, στο κεφάλαιο συγγνώμη, βιώσιμης ανάπτυξης. Περιβάλλον τώρα. Μεγάλη ιστορία. Θα προσπαθήσω να τη συντομεύσω. Το Βιετνάμ αποδίδει μέγιστη προσοχή στην ε, προστασία του περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα τη οικονομικής ανάπτυξης. Υπάρχει περιβαλλοντικό δίκαιο. Το εγκρίναμε από το 1993. Και το 2012 ο Πρωθυπουργό ξεκίνησε τη στρατηγική πράσινη ανάπτυξη και συγκεκριμένο σχέδιο δράση οικολογικό γκρίθηκε. Το 2016, φαντάζομαι το γνωρίζετε, όπως και άλλες χώρες, εγκρίναμε κι εμείς την Συμφωνία των Παρισίων. Με τη Συμφωνία Ελευθερών Εμπορίου θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Έχουμε το κεφάλαιο 13 της Συμφωνίας Εμπορίου. Βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό το κεφάλαιο θα φροντίσει το εμπόριο να μην επιβαρύνει το περιβάλλον, να μην είναι σε βάρος προστασίας του περιβάλλοντος. Δεσμευόμαστε στο προς το Αποτελεσματικά να υλοποιήσουμε τις συμφωνίες πολυμερούς πλαισίου τις οποίες, για το περιβάλλον, τις οποίες έχουμε αναλάβει και για την κλιματική αλλαγή μετά από τη Συμφωνία των Παρισιών και για τα ε, είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και για τη βιοπικιλότητα. Επίσης, δεν θα θυσιάσουμε τα περιβαλλοντικά πρότυπα για να προσελκύσουμε εμπόρου και επενδύσει. Έχουμε αναλάβει σχετική δέσμευση. Το ίδιο και στο πλαίσιο της CPTPP. Αυτό δείχνει τη μεγάλη αποφασιστικότητα της κυβέρνησής μου και τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος. Έρχομαι τώρα στην ε, παράνομη λοτομία και το VPA. Τεθρωτική αυτή συμφωνία. Εμεί θέλουμε να την καταπολεμήσουμε την παράνομη λοτομία. Γι' αυτό είμαστε και από τι πολύ λίγε χώρε περιοχή που συμφωνήσαμε να διαπραγματευτούμε ε, και να ε, προσυπογράψουμε το FLECT και το, το VPA, τη σχετική συμφωνία. Αυτό δείχνει ότι είμαστε αποφασισμένοι να πούμε όχι στην παράνομη ξυλία. Και ελπίζω με την αύξηση τη ευαισθητοποίηση τη επιχειρηματική κοινότητα στο Βιετνάμ και με τι προσπάθειε τη κυβέρνηση και μέσω τη υλοποίηση αυτή τη συμφωνία VPA που θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στι Βρυξέλλε. Ελπίζω λοιπόν ότι σύντομα θα έχουμε θαρρυντικά αποτελέσματα. Τέλος, ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλά είπατε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιβεβαιώνω, κύριε Κέρτον Ντάρλινγκ πως στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης των ΠΟΕ δεν θυμάμαι να αναλάβαμε κάποια δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί ο ΠΟΕ δεν αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διορθώστε να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι αναλάβαμε κάποια τέτοια δέσμευση. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτή τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ, αυτή η συμφωνία εντάσσεται σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο συνεργασία μεταξύ Βιετνάμ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάσσεται, επαναλαμβάνω, σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Επομένω, περιμένουμε να συνεισφέρει στην ενίσχυση των σχέσεων σε όλα τα μέτωπα. Η παρελθούσα εμπειρία στο Βιετνάμ μας δείχνει ότι το εμπόριο και επενδύσεις έχουν εισφέρει τα μάλα στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και στην κοινωνική πρόοδο του Βετνάμ. Εντάσσονται στους στρατηγικούς λόγους για τους οποίους όλα αυτά ε, γιατί έχουμε αυτό το τόσο φιλόδοξο θεματολόγιο που περιλαμβάνει κανόνες για τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα και την ισχυρή συμμετοχή των διπλεκομένων φορέων. Εγώ είμαι ένας ταπεινός εμπορικός διαπραγματευτής. Απλά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είναι εκτός της δικής μου αρμοδιότητας και της δικής μου τεχνογνωσίας άλλοι συνάδελφοί μου στο Βιετνάμ και ομόλογοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πρέσβης που είναι παρόν. Ε, ελπίζω ότι έχουν να σας πούν μια εξαιρετική ιστορία, ακριβώς χάρη στη συνεργασία μας και χάρη στη συμφωνία ε, που έχουμε επιτύχει. Ε, αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ε, και αν μάλλον ξέχασα να απαντήσω, ζητώ συγγνώμη σε κάτι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φυπουργέ που απαντήσατε στα ερωτήματα των βουλευτών. Ολοκληρώθηκε λοιπόν εδώ το πρώτο τμήμα της ακρόασης αυτής και έχουμε για το δεύτερο τμήμα πέντε εμπειρογνώμονες ε, για την Συμφωνία Ελεύθερου Μπορείου με το Βιετνάμ. Καθένας ε, από τελείως διαφορετικό υπόβαθρο. Ελπίζω να είναι και πέντε εδώ ε, για να συζητήσουμε ανοιχτά Νικολά Οντιέ, συμπρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Εμπειρικού Επιμελητηρίου στο Βιετνάμ. Έξι λεπτά το πολύ παρακαλώ. Uh, Έξι λεπτά. Εγώ νόμιζα ότι είχα δέκα λεπτά. Εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ Εισηγητά. Ε, κύριε Υπουργέ, κύριε Κιόνινγκ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είμαι σήμερα εδώ ε, εκπροσωπώντας ε, το ε, Eurocham, ε, το οποίο δημιουργήθηκε το 1998 με 60 μέτρα. Να σας πω ε, ότι εδώ και 30 χρόνια ασχολούμαι ε, με τα νομικά ζητήματα τα οποία απορρέουν από τον ΔΟΕ ε, και σας ε, βεβαιώ ότι η επικύρωση των συνθήκων θα γίνει το 19 με 20. Δύο τρίτα των ε, μελών μας ε, είναι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το πρωί είμαστε στο άλλο κτίριο στην Ολομέλεια που έγινε αυτή η διάσκεψη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ποιοι είμαστε. Η Eurocham δεν χρηματοδοτείται από τις Βρυξέλλες, δεν χρηματοδοτούμαστε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε ακόμα και από την κυβέρνηση το, του Βιετνάμ ή από τον Υπουργό Εμπορίου που μίλησε προηγουμένως. Ε, Αυτό χρηματοδοτούμαστε. και από τα χίλια ε, μέλη μας. Θέλουμε το Βιετνάμ να γίνει μια χώρα φιλική. Ε, θέλουμε ε, ε, ελεύθερο εμπόριο και αυτό κάνουμε εδώ και τόσα χρόνια. Είμαστε τώρα η φωνή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στο Βιετνάμ. Έχουμε 16 sector committees που καλύπτουν πάρα, πολλές, πάρα πολλούς τομείς. Είμαστε λοιπόν ε, η φωνή όλων αυτών των ε, κλάδων από, τον, από την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι τον Ίνο και τα είναι ο πνευματόδη. Εμείς ε, δουλεύουμε σε ολόκληρο το Βιετνάμ, όχι μονάχα στο Ανόη, αλλά και στην ε, ε, Ήπεθρο. Οι κλωστοϊφαντουργίες δεν είναι στο Ανόη ή στις μεγάλες πόλεις, είναι στην Ήπεθρο. Και μάλιστα έχουμε και στην Χαϊφόν, τη δεύτερη μεγάλη πόλη, και πολύ σημαντική ε, περιφέρεια στην, στο Βιετνάμ έχουμε οπωσδήποτε και εκεί ε, γραφείο. Είμαστε λοιπόν ε, δραστήριοι και δραστηριοποιούμε σε ολόκληρο το Βιετνάμ. Επίσης, Έχουμε και εκπροσώπηση ε, στην περιφέρεια ε, η οποία επικεντρώνει την μεγαλύτερη δραστηριότητα για την κλωστοϊφαντουργία και τα είδη ένδυσης υπόδησης. Ε, να σας πω ότι δύο φορές ε, τον χρόνο. Εμείς δημοσιεύουμε την Λευκή Βίβλο πάντα σε ε, αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο ε, Εμπορίου. Ευχαριστούμε κύριε Χάνα, καθώς επίσης και με το Υπουργείο που ασχολείται και είναι υπεύθυνο με τις επενδύσεις. Σας ξαναλέω, είμαστε η φωνή του Βιετνάμ ως Eurocham και θέλουμε ε, μέσω της Eurocham ε, να προωθήσουμε τις αρχές για τις αξίες του ελεύθερου εμπορίου έτσι όπως εμείς τις πρεσβεύουμε στην Ευρώπη. Τα τελευταία 30 χρόνια είμαι στο Βιετνάμ και να σας πω ότι είναι μια τρομερή χώρα. το 1987 αποφάσισε ε, το Βιετνάμ να ανοίξει τα σύνορά του στις ξένες ε, επιχειρήσεις ε, και μέσα σε μερικά χρόνια άλλαξε η κατάσταση. 6% ο ρυθμός ανάπτυξης κάθε χρόνο. Όταν ε, πήγα στο Βιετνάμ, δύο δολάρια τη μέρα ε, είχε ο κάθε πολίτης. Ε, τώρα αυτό έχει αλλάξει. Όταν πήγα στο Βιετνάμ, 50% των σπιτιών στο, δεν είχαν πρόσβαση στο ηλεκτρικό. Τώρα σε όλα τα χωριά, στο βορρά, στο νότο του Βιετνάμ, Πάντα υπάρχει και παντού ε, ηλεκτρισμός, πάντα ε, βλέπεις ότι τα παιδιά πηγαίνουν ε, σχολεία, πολύ συχνά πηγαίνουν τα παιδιά και στο Χανόι για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Όσον αφορά το ΑΕΠ, από 400 δολάρια έφτασε στα 2.000 δολάρια. Ε, επομένως, τα τελευταία 30 χρόνια, τελευταία 30 χρόνια επενδύσεων και δραστηριοτήτων ε, ε, στην, στο Βιετνάμ τα πράγματα προχώρησαν. Θα ξέρετε, φαντάζομαι, ότι το Βιετνάμ έχει 16 διμερείς συμφωνίες. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθα σε επαφή με τον ε, Πρωθυπουργό, ο οποίος θα έρθει μάλιστα και στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα. Και ε, πρέπει να σας πω ότι η Samsung, ας πούμε, επενδύει στην, ε, στο Βιετνάμ σχεδόν όσο επενδύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης να σας πω ότι το Κορεατικό Επιμελητήριο έχει 10.000 μέλη γιατί είναι πάρα πολλοί οι Κορεάτες οι οποίοι ζουν και επενδύουν στο Βιετνάμ. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ε, είπε ε, ε, και ο Πρωθυπουργός της Κορέας είπε ανοίξτε τα σύνορά σας ε, στις ε, επενδύσεις γιατί και εμείς θα επενδύσουμε στην χώρα σας. Από την άλλη πλευρά δεν είναι μόνο η Κορέα που επενδύει, επενδύει και η Κίνα. Αυτή η One Belt One Road Policy έχει ξεκινήσει ε, στην, ε, στο Βιετνάμ. Ε, πραγματικά σας λέω, υπάρχουν σύνορα με, με το Βιετνάμ και αυτή η πολιτική One Road, One Belt ισχύει. Επομένως η Κορέα είναι στο Βιετνάμ, η Κίνα επενδύει και είναι στο Βιετνάμ. Επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στο Βιετνάμ. Α, ναι, δεν έχω χρόνο, ε, τι κρίμα. Να σας πω πριν τελειώσω ότι δουλεύουμε από το 2012 για, το, ε, για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με το ε, Υπουργείο Εμπορίου ως Eurocham. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και για το follow-up και την λεγόμενη gap ανάλυσης. Εδώ έχουμε την έκθεση για το θέμα αυτό και θα τα δώσω στους φίλους ε, εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσατε να εκλεγείτε βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το λόγο που είχατε. Θα προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Κάρον Κιόρτης, είναι από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και θα μα μιλήσει για την άποψη αυτού του οργανισμού για την Συμφωνία Ελευθερών Εμπορίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ΔΟΕ θα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση σε αυτή τη συζήτηση. Θα σας παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο η ΔΟΕ βλέπει αυτή την ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου από την πλευρά του διεθνού Οργανισμού εργασία, από την πλευρά των δικών μα αρχών. Ε, είναι προφανέ ότι όλοι γνωρίζετε τον ΔΟΕ, φάνηκε από τι ερωτήσει αυτό, ε, γνωρίζετε και τι συμβάσει του, ίσως όμω να μην γνωρίζετε με ποιον τρόπο έχει εμπλακεί, έχει συνεργαστεί ο ΔΟΕ με το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ έγινε μέλο του το 1992 από τότε. Σταδιακά έχει επικυρώσει τις συμβάσεις του Ανοίξαμε γραφεία το 2003 στη χώρα και από τότε παρακολουθούμε και συνεργαζόμαστε με τη Βιτνάμεζικη κυβέρνηση για την επικύρωση αυτών των συνθήκων και για την εφαρμογή τους στην πράξη, ε, την εφαρμογή στην πράξη των εθελοντικών δεσμεύσεων του. Πέντε από τις οχτώ κύρια συμβάσεις του ΔΟΕ έχουν επικυρώσει το Βιετνάμ. Αυτό είναι ο μέσος όρος της χωρών της περιοχής έχει επίσης εκφράσει την επιθυμία του να επικυρώσει τις άλλες τρεις. Αυτό θα έλεγα είναι ότι ε, σπάνιο και θετικό για την περιοχή. Το που παραμένει είναι τα ζητήματα τα υγειονομικά και βεβαίω τα ζητήματα των εργαζομένων στη θάλασσα. Όπω έλεγε και ο Υφυπουργό προηγουμένω, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση του Βιετνάμ στην μεταρρυθμίση του εθνικού του δικαίου μετά την επικύρωση αλλά επίσης να προωθήσουμε και την επικύρωση και άλλων διεθνών προτύπων που σχετίζονται με τις κύριες αυτές συμβάσεις. Η Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ θα δώσει τη δυνατότητα στον ILO να συνεργαστεί περισσότερο με την κυβέρνηση του Βιετνάμ προ αυτή την κατεύθυνση, όσον αφορά τώρα τη μεταρρύθμιση του, του εργατικού δικαίου έχουμε υποστηρίξει επί χρόνια την μεταρρύθμιση και την αλλαγή του εργατικού δικαίου έτσι ώστε να, έρθει, να γίνει συμβατό με τα διεθνή πρότυπα. Έχουμε συνεργαστεί με τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου σε συνεργασία μάλλον με τους κοινωνικούς εταίρους έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό και έτσι ώστε να εφαρμοστεί και στην πράξη. Συνεργαζόμαστε επίσης με την κυβέρνηση του Βιετνάμ για να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο ε, σχέσεων εργοδοτών εργαζομένων που να πληρεί περισσότερο τις διεθνείς προδιαγραφές για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να δημιουργηθούν οι τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τη δημιουργία εκλεγμένων συνδικαλιστών εκπροσώπων των εργαζομένων στις διάφορες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη και καλύτερη αντιπροσώπευση και των οργανώσεων των εργοδοτών και των οργανώσεων των ε, εργαζομένων. Έχουμε κάνει επίσης μια αξιολόγηση του αντικτύπου αυτών των μεταρρυθμίσεων και των τριμερών διαπραγματεύσεων. Επίσης, ο ILO δραστηριοποιείται στο Βιετνάμ προωθώντας αυτά τα ζητήματα και στο επίπεδο των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταπίσης τροφίμων. Έχουμε τρεις βασικούς στρατηγικούς στόχους. Πρώτον, να υποστηρίξουμε την προσπάθεια του Βιετνάμ να ενταχθεί στο διεθνές γίγνεσθε. Δεύτερον, να προωθηθεί ε, να προ... Είναι το ζήτημα λοιπόν του θεσμικού πλαισίου για τις εργασιακές σχέσεις. Η ανάπτυξή του στι επιχειρήσει, καθώς επίση και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό που στην Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου εντάσσονται και ζητήματα τέτοια ε, εργατικού δικαίου. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνει κατάπτυση στην εφαρμογή των διεθνών προτύπων. Ε, υπενθυμίζεται επίση το γεγονό ότι τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ολόκληρο το Βιετνάμ, χωρί να υπάρχουν κάποιε ζώνε ειδικού οικονομικού ενδιαφέροντο όπου να αποκλείονται. Όπω ανέφερε πριν και ο Υφυπουργό και άλλοι συνάδελφοι πριν. Υπάρχει ένα σοδικό χάρτη από την κυβέρνηση του Βιετνάμ, έτσι ώστε να εφαρμόσει τους στόχους της διακήρυξη που έκανε το 1999. Αυτό σημαίνει αναθεώρηση του εργατικού κώδικα που είναι απαραίτητο για να μπορέσουν το Βιετνάμ να ακυρώσει και τις υπόλοιπες συμφωνίες του ΔΟΕ. Του χρόνου προβλέπεται να εγκριθεί αυτός ο νέος κώδικας εργατικού δικαίου στο Βιετνάμ, όπως μας έλεγε και ο Φουπουργό, και αυτό θα ανοίξει το δρόμο για την κύρωση της Σύμβασης 98, η οποία προσπαθεί να καταπολεμήσει την επέμβαση των εργοδοτών στα, στην εκπροσώπηση των εργαζομένων και ανοίγει το δρόμο για ουσιαστικές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Βλέπουμε ότι προοδευτικά λοιπόν υιοθετούνται οι συμβάσεις του ΔΟΕ. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση του Βιετνάμ προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε διάφορα προγράμματα στη χώρα και ορισμένα από αυτά χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα συγκεκριμένο μάλιστα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας και την πρόθεση των υπολείπων συμβάσεων του ΔΟΕ. Μας βοηθούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την προσπάθεια. Το κεφάλαιο της ε, Συμφωνίας Ελευθέρων Εμπορίου νομίζω θα βοηθήσει στην πολιτική δυναμική έτσι ώστε να υιοθετηθούν αυτά τα πρότυπα. Εάν το Βιετνάμ και άλλε χώρε υιοθετήσουν και τι υπόλοιπε συμβάσει, αυτό συνεισφέρει γενικότερα στο να υιοθετηθούν από πολλέ άλλε χώρε. Ο ΔΟΕ θεωρεί ότι η κυβέρνηση του Βιετνάμ έχει αντιληφθεί ότι δεν ε, μπορεί να υπάρξει μια ε, καλύτερη θέση στον διεθνή ανταγωνισμό με το να παραγνωρίζονται τα εργατικά δικαιώματα. Ευχαριστώ και τώρα τον κύριο Γκραν, ειδικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ. Μεγάλη χαρά που τον καλωσορίζω και του δίνω το λόγο να μα πει τι απόψει του. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε και κύριοι, σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην ακρόαση αυτή. Θα περιοριστώ σήμερα μόνο στον εκδημοκρατισμό των ανθρώπινων δικαιώματα και στο πώς σχετίζονται με την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Πρώτα απ' όλα, δύο πράγματα, δύο γεγονότα θέλω να αναφέρω και θα κάνω μετά πέντε παρατηρήσεις καταλήγοντας δε με τρεις συστάσεις. Πρώτον, το πρώτο γεγονός. Uh, το κείμενο της Συμφωνίας Εύθος των Αλλαγών έχει εγκριθεί μετά από μακρύς διαπραγματεύσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Βιετνάμ. Δεύτερον, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ είναι κακή και επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια. Παρατήρηση. Πρώτη. Υπάρχουν ενδείξεις αρκετές ότι με τη δημοκρατία ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα βελτιώνονται. Και μάλλον με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν θα δείξουμε πώς μπορούμε να αντλήσουμε πολύ χρήσιμα διδάγματα από γνωστά ιστορικά και εμπειρικά μαθήματα επιτυχούς εκδημοκρατισμού. Πρώτη λοιπόν παρατήρηση είναι, μελέτες εξυγχρονισμού ξεκάθαρα δείχνουν ότι οι διαδικασίε εξυγχρονισμού δημιουργούν ευνοϊκές διαρθρωτικές συνθήκες για εκδημοκρατισμό και παγίωση εδραίωση νέων δημοκρατιών. Δεύτερον, η αποτελεσματικός, ο αποτελεσματικός εκδημοκρατισμός Χρειάζεται και ένα επιτυχημένο κοινωνικό κίνημα. Χρειάζεται δηλαδή μία κοινωνία πολιτών που να είναι ζωντανή και που να προωθεί την ανέλυξη του ανθρώπου. Η Συμφωνία Ελευθερομπορίου και το TPP και το CPTPP απαιτούν από το Βιετνάμ να να ακυρώσει τις βασικές συμβάσεις της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 87, 98 και 105. Όλες αυτές έχουν επίπτωση στην κατάσταση και την ανάπτυξη των δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο μπορεί να γνωρίζουν πώ επηρέασαν οι συμφωνίες του Ελσίνκη του 1975 την ανάπτυξη της ε, κοινωνίας των πολιτών στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στη δεκαετία του 80. Ξέρουμε πόσο σημαντικά συνεισέφεραν στη δημοκρατική μετάβαση στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη ότι προώθησαν τον εκδημοκρατισμό το 1989. Δεν εστιάζει μεν στα ανθρωπινά δικαιώματα, δημοκρατία, η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, όπως όμως και οι συμφωνίες του Ελσίν και έτσι και η Συμφωνία Ελεύθερου θα επηρεάσει αντίστοιχα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό του Βιετνάμ. Τέταρτη παρατήρηση. Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου θα επηρεάσει θετικά τα οικονομικά δικαιώματα των Βιετναμέζων. και αυτά θεωρούνται ανθρώπινα. Είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Πέμπτη παρατήρηση. Γενικώ είναι αποδεκτό από τους ε, επιστήμονες, από τους ακαδημικούς, ότι η ένταξη στην παγκόσμια αγορά αυξάνει και την επιρροή της διεθνού πίεση. Αν κυρωθεί η Συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μεγαλύτερε δυνατότητες ε, άσκησης πίεσης ε, στο Βιετνάμ σε μελλοντικέ διαπραγματεύσεις. Αυτές οι παρατηρήσεις συνεπάγονται και ένα σημαντικό γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό στοιχείο το οποίο δεν ανέφερα ότι μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί η εξάρτηση του Βιετνάμ από τον ισχυρό γείτονα. Και έρχομαι στις συστάσεις μου. Και αυτά τα πέντε διδάγματα, οι πέντε αυτές παρατηρήσεις, νομίζω στηρίζουν την επικύρωση της Συμφωνίας Δευτεροπορίου, επομένω ποιε είναι οι τρεις μου συστάσεις. Πρώτον, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει, να διασφαλίσει ότι το Βιετνάμ θα υπογράψει και θα κυρώσει τις τρεις ε, βασικές συμβάσεις της Διεθνής Οργανωσίας και με τα χαράς άκουσα ότι αυτό είναι το σχέδιο της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το TPP συμφωνία μεταξύ Βιετνάμ Ηνωμένων Πολιτειών ήταν πολύ πιο ισχυρή από την σκύρωση της σύμβασης του, της ΔΟΕ. Υπάρχει και η δήλωση από τις 7 Οκτωβρίου που λέει ότι θα κυρώσει ο Πρωθυπουργό τις επόμενες εβδομάδες του CPTPP. Βιετνάμ και η Ιαπωνία έχουν ζητήσει από τη είπα να επανέλθουν στο TPP. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει το Βιετνάμ να κυρώσει τη συμφωνία και ότι μάλλον θα επιτύχει σε αυτή την προσπάθεια. 6 Αυγούστου φέτος στήσαμε από την Εθνοσυνέλευση του Βιετνάμ να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν Πόσο μάλλον το καλύτερο θα ήταν να γίνει αυτόν τον Οκτώβριο. Δεύτερο, δεύτερη σύσταση. θα πρέπει ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, οι οργανώσεις των πολιτών να είναι ανεξάρτητε και να ενταχθούν στους μηχανισμού παρακολούθησης τη συμφωνίας. Όπως εμπόριο βιώσιμη ανάπτυξη, το TSD και DAG, που είναι οι εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες. Τρίτη σύσταση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο μηχανισμό να ε, θεσπίσει ή να βελτιώσει τους μηχανισμούς του άρθρου Χ 17 παράγραφος 2 της Συμφωνίας Ελευθερμπορίου και το άρθρο 57 PCA. Ώστε αν δεν τηρήσει τις συμφωνίες του Βιετνάμ στο πλαίσιο της PCA να μπορεί να υπάρξει αναστολή Τη Συμφωνία Ελεύθερου Μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρετε αυτό. Είναι εύκολο για εσά. Αν λοιπόν αυτέ οι συστάσεις εκπληρωθούν, θα νιώθει πάρα πολύ πιο έτοιμη η ανεξάρτητη κοινότητα κοινωνία των πολιτών στο Βιετνάμ να υποστηρίξει αυτή τη συμφωνία. Τέλος, θέλω να αναφέρω την περίπτωση ενό πολιτικού κρατουμένου στο Βιετνάμ. Νομίζω ότι πρέπει να απελευθερωθεί ε, όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, ε, αλλά θα αναφέρω συγκεκριμένα τον Τραν Χουν Ντουι Τουκ, ε, που είναι αντιρρησία συνείδηση και πρόσφατα σε επιστολέ του από τη φυλακή ένα επιτυχημένο ε, επιχειρηματία, ο Τραν Χουν Ντουι εξέφρασε την υποστήριξή του για το Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Είπε ότι είναι μια ευκαιρία για να προχωρήσει πολύ γρήγορα ο ξεχωρισμός του Βιετνάμ και να μειωθεί οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση για το Βιετνάμ από τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΙΠΑ Κίνας. Έχει δεκτεί στα 9 από τα 16 χρόνια κάθριξης που το έχει επιβληθεί. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη χρονική στιγμή για να τον απελευθερώσει η Βετναμέζικη κυβέρνηση από τώρα. Αυτόν τον Τουκ, τον υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον υπερασπιστή του ελεύθερου εμπορίου. Είναι ένα μεγάλο ατού για τη χώρα. Δεν πρέπει να σαπίζει στη φυλακή. Του ζήτησαν οι αρχές να ομολογήσει για να μπορέσει να απελευθερωθεί. είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς πρέπει να σας διακόψω, λέει ο κύριος Λάγκε. Λυπούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι αντιμετωπίσατε προβλήματα για να φτάσετε εδώ, όμως νομίζω το μήνυμα έγινε σαφές παρόλα αυτά και σας ευχαριστούμε πολύ. Ms. Anja von Molke, Trade Hub Unit. Έχουμε μαζί μας και το, την επικεφαλή του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, λέει η κυρία Βον Μόλτκε. Η περιβαλλοντική πτυχή των, ε, του θεματολογίου για την βιώσιμη ανάπτυξη ε, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ θα μιλήσω για τη σχέση περιβάλλοντος ε, και ε, εμπορίου, καθώς επίσης και τις περιβαλλοντικές διατάξεις εντός των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου FTAs και την ιδιαίτερη κατάσταση στο Βιετνάμα, καθώς επίσης και την δυνατότητα χρήσης της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου για το περιβάλλον. Πρώτα απ' όλα, στόχος ε, του Environment and Trade Hub ε, είναι να ε, βελτιώσει την διασύνδεση ανάμεσα στο εμπόριο και την διακυβέρνηση και τις περιβαλλοντικές πολιτικές, πάντα στα πλαίσια των πεδίων εστίασης, ε, περιβάλλον, ε, σωστές τεχνολογίες, δημιουργία αλυσίδας αξίας και ε, ελάφρυνση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ήδη ακούσαμε ότι η απελευθέρωση του εμπορίου εξορισμού προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και ένα διαφορετικό μείγμα οικονομικών δραστηριοτήτων που όμως μπορεί να αυξήσουν την πίεση ε, προς το περιβάλλον. Για αυτό λοιπόν εντός των FTA εμείς ε, ε, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ελαχιστοποιείται η πίεση στο περιβάλλον και ότι χρησιμοποιείται σαν ένα θετικό ε, στοιχείο περιβαλλοντικής πολιτικής, αυξάνοντας τα επίπεδα περιβαλλοντικής ευαισθησίας ε, της ε, χώρας και εντασσόμενη βεβαίως σε, σε δυνατότητες προστασίας, στην ικανότητα προστασίας του περιβάλλοντος μέσω συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων και πολιτικών. Ε, μας ενδιαφέρει να γίνει κατανοητή η διασύνδεση ε, ανάμεσα στην ε, γνώση και την κατανόηση την από και από την, και την διαπραγμάτευση και την υλοποίηση από την άλλη. Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε διατάξεις μέσω των οποίων προωθούνται υπερβολοντικοί στόχοι και σκοποί. οι ίδιες οι περιβαλλοντικές ε, διατάξεις ε, μπορούν να εφαρμοστούν από μόνες τους, αλλά έχουν καλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον εάν ενταχθούν ε, στις εμπορικές συμφωνίες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι το περιβάλλον αποτελούν πολύ σημαντικό τμήμα, κομμάτι των FTAs, 85% των FTAs πλέον περιλαμβάνουν ε, κάποια, ε, κάποιες περιβαλλοντικές ε, ρήτρες. Στην δε προκείμενη περίπτωση, σε γενικές γραμμές, ναι, μπορούμε να πούμε ότι κάθε συμφωνία έχει περίπου 60 διαφορετικά είδη περιβαλλοντικών διατάξεων. Στο Βιετνάμ βλέπουμε έχουμε ένα εξαιρετικά διαφοροποιημένο πεδίο, μια χώρα πολύ διαφοροποιημένη. Ε, έχουμε στο Βιετνάμ περίπου 10% ε, της ε, χλωρίδας και της επανίδας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη περιβαλλοντικά, ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, κυρίως όσον αφορά την άνοδο του επίπεδου της θαλάσσης. Ε, γι' αυτό ε, έχουν ληφθεί ιδιαίτερα, ε, ιδιαίτερη να έχει ληφθεί όσον αφορά την θωράκιση της χώρας και απέναντι στην την διαχείριση των αποβλήτων, την χρήση χημικών, κυρίως απέναντι δηλαδή στις στην εκβιομηχάνηση της ε, χώρας ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ε, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα αμβλύνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Χάν που αναφέρθηκε ακριβώς στην μεταρρύθμιση την νομοθετική ε, το, το Βιετνάμ είναι ε, από τις ε, πρώτες χώρες που έχει δημιουργήσει ένα σύστημα για, την, για τη μόλυνση. Επίσης, το Βιετνάμ έχει επικυρώσει πολλές περιβαλλοντικές συνθήκες και συμβάσεις, αλλά εδώ θα ήθελα να πω ότι το κύριο διακύβευμα και η μεγάλη πρόκληση είναι βέβαια ε, η, ε, η υλοποίηση, η εφαρμογή. Ε, είναι ε, ε, λιγότερες οι λιγότερες οικονομικές δυνατότητες που δίνονται όσον αφορά την υλοποίηση. Ε, για να επανέλθω στην διασύνδεση ανάμεσα στους στόχους του περιβάλλοντος και του ε, ε, εμπορίου ε, να σας πω ότι έχει γίνει πριν μερικά χρόνια μελέτη αντικτύπου για τις χώρες Ασεάνα αλλά πολλά από τα ευρήματα μπορούν να εφαρμοστούν και να ισχύσουν και για την προκείμενη περίπτωση και επομένως γνωρίζομαι ότι ε, υπάρχουν οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε υπεραλίευση, ε, σε περιβαλλοντική ε, μόλυνση. 80% των ασθενειών στο Βιετνάμ προέρχονται από την μόλυνση των υδάτων. Επομένως θα πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί στο Βιετνάμ που ε, θα υποστηριχθούν και θα αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα και τα προβλήματα. Επίσης ε, είναι ε, σημαντικό να δούμε τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου σαν περιβαλλοντικά εργαλεία, σαν δυνατότητες για περαιτέρω capacity building. Δεν θα αναφερθώ στις διατάξεις, δεν έχουμε το χρόνο. Ωστόσο, να σας πω ότι ε, η Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή ευκαιρία έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δουλέψει σε στενή συνεργασία με το Βιετνάμ έτσι ώστε να δημιουργηθεί πράσινη οικονομία, πράσινες θέσεις ε, εργασίας, ε, να αποφευχθεί η αρνητική επίπτωση που μπορεί να έχουν οι ενισχυμένες οικονομικές δραστηριότητες και ε, για να δημιουργηθεί μια, ένα σωστός διάλογος μεταξύ όλων των τμήματων της οικονομίας. Ε, τέλος, όσον αφορά τις συστάσεις, τεχνική αρρωγή, δυνατότητα ε, οικοδόμησης ε, ικανοτήτων, ε, υλοποίηση όλων των προσδοκόμενων στόχων, γιατί όλες οι διατάξεις το που αφορούν την ε, βιώσιμη ανάπτυξη ε, είναι προσδοκίες και ευκταία και όχι υποχρεωτικές ε, διατάξεις. Και τέλος, η επιτήρηση της βιωσιμότητας όλων των δραστηριοτήτων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, να σας πούμε από πλευρά του Τμήματος Περιβάλλοντος Εμένων Εθνών ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Τελευταία ομιλήτρια, κυρία Λεωνόρα Κατέλα, ε, σύμβουλος στην Business Europe. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση που δίνετε την δυνατότητα στον οργανισμό μας, την Business Europe, να σας παρουσιάσει τη θέση της, τις απόψεις της, για την Συμφωνία Ελευθέρων Πορείων με το Βιετνάμ. Η οργανισμό μας εκπροσωπεί τους εργοδότες σε 34 χώρες, μικρών, μεγάλων, μεσαίων επιχειρήσεων. Προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση προς την κατεύθυνση της, του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης στην Ευρώπη, επομένως υποστηρίζουμε το ελεύθερο εμπόριο, ε, υποστηρίζουμε την φιλόδοξη ε, ατζέντα για το ελεύθερο εμπόριο που επιδιώκει η Επιτροπή τα τελευταία χρόνια και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών. Για τρεις λόγους οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υποστηρίζουν αυτήν τη συμφωνία. Οι δύο είναι κου χαρακτήρα και οικονομικού χαρακτήρα και ο τρίτος είναι ο χαρακτήρας, ο ίδιος ο χαρακτήρας της συμφωνίας. Πρώτα απ' όλα, ένας από τους πρώτους λόγους για να υποστηρίζουμε αυτήν την συμφωνία είναι η στρατηγική της διάσταση. Πρόκειται για μια περίοδο όπου το ελεύθερο εμπόριο ε, αμφισβητείται, ότι υιοθετούνται προστατευτικές πολιτικές. Επομένως, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να ενισχύσει τους δεσμούς που έχει με την περιοχή της νοτιοανατολικής αξίας. Μια περιοχή δυναμική που αναπτύσσεται γρήγορα. Το Βιετνάμ ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι μια χώρα που επίσης αναπτύσσεται γρήγορα, έχει 100 εκατομμύρια ε, πληθυσμό, έχει σταθερή ε, θετική ανάπτυξη τα τελευταία 6 χρόνια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης πέρυσι ήταν 6,8%. Είναι εντυπωσιακό αυτό το νούμερο. Είναι η πρώτη τέτοιου τύπου συμφωνία που συνάπτεται με μια αναπτυσσόμενη χώρα και θα έλεγα ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα για άλλες συμφωνίες με άλλες χώρες, καθώς επίσης και ως ε, στοιχείο ε, το οποίο θα οδηγήσει σε μια συμφωνία region to region, από τη μια ε, πολυμερή συμφωνία μεταξύ πολλών χωρών με πολλές χώρες που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ εμείς προτιμούμε αυτές, αυτή τη μορφή συμφωνιών. Γιατί θεωρούμε ότι αυτές οι συμφωνίες ανοίγουν μεγαλύτερες ευκαιρίες, περισσότερες ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις ιδιαίτερα, που θα με τη διευκόλυνση που τους δίνεται να είναι πιο ξεκάθαρο το ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεύτερος λόγος. Είναι επειδή θεωρούμε ότι αυτές οι συμφωνίες ελευθέρων εμπορίου είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από άλλες περιοχές, από επιχειρήσεις από άλλες περιοχές του κόσμου, επειδή ακριβώς το Βιετνάμ έχει συνάψει συμφορίες ελευθερων εμπορίου και με άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι η πολιτική του. Επομένω, θα ήταν δυσμενές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να καθυστερήσουν και να φτάσουν αργότερα από τις υπόλοιπες ε, χώρες και ακόμα χειρότερο να μην υπάρξει καν συμφωνία. Κάθε κεφάλαιο έχει πλέον εκτήματα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δεν θα αναφερθώ σε όλα, αλλά στα πιο σημαντικά. Πρώτα απ' όλα υποστηρίζουμε το εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο για τους ε, απελευθέρωση των δασμών. Ε, ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε ξαφνικές αυξήσεις των δασμών μέχρι και τις τάξεις του 50% για ορισμένε περι, ε, περιπτώσεις. το Βιετνάμ επίσης είναι και χώρα που εισάγει μάλλον είναι η χώρα από την οποία εισάγουμε. Ε, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν μόνο οι εξαγωγές των προϊόντων μας προς τη χώρα αυτή. Έχουμε και εισαγωγές πρώτων υλών ή μερικώς μεταποιημένων προϊόντων από τη Βιετνάμ προς την Ευρω... τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπου γίνεται η τελική επεξεργασία εδώ. Θα θέλαμε και άλλες χώρες όπου να ήταν εξίσου ανοιχτέ όπως και να το θεωρούν εξίσου σημαντικό όσο το Βιετνάμ να ανοίξουν την αγορά των δημοσίων προμηθειών του. Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες πόλει. αλλά εκτός αυτού υπάρχουν νομοσοκομεία που θα πρέπει να χτιστούν σε πολλέ περιοχές. Ε, το Βιετνάμ βελτιώνει τις υποδομές του. Έτσι λοιπόν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να συμμετάσχουν και σε προκηρύξει για όλα αυτά τα έργα και θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν και τοπική παρουσία. Ε, ε, θα υπάρξουν προκηρύξεις επίσης και για τον τομέα των υπηρεσιών. Ένας πολύ σημαντικός τομέας επίσης θα είναι και οι σιδηρόδρομοι. Μετά, ένα, ένα σημαντικό κεφάλαιο τη συμφωνία για εμά είναι οι, οι δημόσιε επιχειρήσει, οι επιχειρήσει υποκρατικό έλεγχο. Έχει κάνει πολλά το Βιετνάμ για να γίνει ανοιχτή οικονομία, οικονομία τη αγορά, αλλά το κράτος συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό πιστεύουμε εμείς ότι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι το Βιετνάμ η μόνη χώρα στην οποία το κράτος είναι σημαντικό παίκτη στην οικονομία. Ε, είναι πολύ σημαντικό για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να έχουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τις τοπικές επιχειρήσεις, με τις βιετιναμέζικες επιχειρήσεις. Μετά βλέπουμε τις προβλέψεις για το ε, η πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό που ε, εμεί θεωρούμε το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του κεφαλαίου είναι αυτά που προβλέπονται για την εφαρμογή. Και τώρα για το TSD, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχουν πολύ, πολλά υποθεί ε, για τις δεσμεύσει που αναλαμβάνει το Βιετνάμ με ξεκάθαρο οδικό χάρτη. Μπορώ να πω ότι και εγώ η ίδια έχω διαπιστώσει ότι το Βιετνάμ προσπαθεί να καταλάβει η κυβέρνηση του Βιετνάμ προσπαθεί να καταλάβει ποιο θα ήταν ο καλύτερο τρόπο για να εφαρμόσει αυτέ του δεσμεύσει για την βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουν δημιουργηθεί, δημιουργούνται μάλλον αυτέ οι συμβουλευτικέ ομάδε οι οποίε θα παρακολουθούν την εφαρμογή του κεφαλαίου TSD. Παρευρέθη σε μια συνάντηση στην οποία είχαν εκπροσώπους από το Υπουργείο Εργασία, από το Υπουργείο Βιομηχανία και Ανάπτυξη και προσπαθούσαν να αντιληφθούν αυτοί οι εκπρόσωποι των Υπουργείων του Βιετνάμ πώς αντιλαμβάνεται αυτές τις διατάξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τι πρέπει να φτιάξει θεσμικά το Βιετνάμ για να εφαρμοστούν αυτά. Συμπερασματικά, πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει δυνατότητες για ανάπτυξη στο Βιετνάμ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο βιώσιμο και πιστεύω ότι μια τέτοια συμφωνία θα αυξήσει τις πιθανότητες που έχουμε πολύ περισσότερο από το να μην έχουμε συμφωνία, να πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους εμπειρογνώμονες. Μας δώσατε μία πλήρη επισκόπηση της κατάστασης. Πολύ ενδιαφέρουσες επιτυχίες, ε, ελπιδοφόρες για το μέλλον. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση, ολοκληρώθηκε η ακρόαση. Θα δώσω το λόγο στους, ε, στην μάλλον ε, πρόεδρο του Επιτροπής, ε, υποετροπής. Δεν μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Ξέρετε, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Έχετε ερώτηση για κάποιο συγκεκριμένο ομιλητή. Όχι, ωραία. Επόμενο, κύριε Λόχμπίλερ, για να καταλήξουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, ε, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Αυτή τη στιγμή μιλάω ως εισηγήτρια από την ΑΦΕΤ για τη συμφωνία PCA ε με το Βιετνάμ και συγχαίρω θερμά ε, το Βιετνάμ που κατάφερε να έχει αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Πράγματι, εγγυάται το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στα τρόφιμα, στη στέγαση για, τόσα πολλά, για τόσους πολλούς ανθρώπους. Κύριε Υφυπουργέ, βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει αντίφαση. Ε, μπορείτε να βελτιώσετε και τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα και τότε η κατάσταση είναι ακόμη καλύτερη. Οικονομική πρόοδος με κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Τον Ιούνιο ακούσαμε κάποιε θετικέ ε, δηλώσει από τον Υπουργό Εμπορίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά παραμένουν επί χάρτου αυτά μέχρι στιγμή, ε, Άκουσα πολύ προσεκτικά ότι έχετε ένα σχέδιο να εγκρίνετε και τις τρεις ε, απομένουσες συμβάσει του ΔΟΕ μέχρι τον Νοέμβριο το 2019. Ελπίζω να το τηρήσετε αυτό το χρονοδιάγραμμα, θα ήταν καλό. Στοιχώ, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όμω επιδεινώνεται η κατάσταση. Έχουμε πολλέ αντιρρησίε συνήθω στη φυλακή. Πρέπει αυτοί να απελευθερωθούν. Οι, πολιτικοί κρατούμενοι τέλο πάντων πρέπει να απελευθερωθούν. Συστηματικά συλλαμβάνονται ξυλοδαρμού, βλέπουμε βασανιστήρια ε, για τους ανθρώπους οι οποίοι τι έκαναν, απλά άσκησαν την ελευθερία ε, έκφρασης και εκφράστηκαν κατά των δρακόντιων νόμων. Έχουμε επιδείνωση τη κατάσταση δεν ελέγχονται τα επενδυτικά προγράμματα. Αυτό επηρεάζει και τον πληθυσμό στην Ήπεθρο. Το 2016, για παράδειγμα, εκατοντάδες αλείς, χιλιάδες αλείς έχασαν τα προστοζήν. Όταν η Φορμόσα ε, έριξε τοξικά απόβλητα και κιάνιο ε, στη θάλασσα με τεράστιες απώλειες. Ε αναζητούσαν υποζημίωση οι πληγέντες και τους εκφόβησαν για να μην πω ότι τους ε, απείλησαν. Ε, και πολλοί 32 συγκεκριμένα βουλευτές τον προηγούμενο μήνα έγραψαν ε, στην επέτη εκπρόσωπο Μογκερίνη ζητώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει σαφή σημεία αναφορά benchmark για τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν την ε, υλοποίηση συμφωνία. Και η επενδυτική συμφωνία δημιουργεί περισσότερε ανησυχίε σε ό,τι αφορά ε, το σεβασμό του διεθνού ανθρωπίνου δικαίου. Ότι δεν υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης ε, για η επίλυση διαφορών όταν έχουμε τι επενδύσει να επηρεάζουν αρνητικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει αλληλευκό εξοδότηση για παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να υπάρξει ένα πρωτόκολλο και μια ερμηνευτική δήλωση, διακήρυξη που θα προσαρτηθεί στη συμφωνία που θα λέει ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων κοινωνίας των πολιτών και θα πρέπει να έχουμε και ένα μηχανισμό επίλυσης προβλημάτων όταν, για παράδειγμα, οι επενδύσεις επηρεάζουν αρνητικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι βέβαια όταν προσκαλούνται οι ΜΚΟ θα, να κάνουν κάτι θα πρέπει να το κάνουν χωρίς φόβο και ελεύθερα. Ελπίζω να πάρετε μαζί σας το μήνυμα, το μεταφέρετε στην πατρίδα σας σε ό,τι στην Επιτροπή για, τις, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς σχέσεις. Και ελπίζω να υπάρξει βελτίωση. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο νέος πρόσβησε του Βιετνάμ πολύ σύντομα. Πόσα, χρή, πόσα λεπτά έχω γιατί θέλω να απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις. Μπορώ να έχω πέντε λεπτά. Πρέπει να σταματήσουμε ακριβώς και μισή. Βεβαίως ξέρετε ότι μπορούν να γίνουν διμερείς επαφές μετά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία λοιπόν. Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ε, τέλεια η κατάσταση στο Βιετνάμ. Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε δηλαδή μια ισορροπημένη προσέγγιση ε, και να αναγνωρίσει κανείς τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που παρουσιάζει η κατάσταση με τα Ηνωμένα Έθνη έχουμε συζητήσει πολλά θέματα. Να σας πω λοιπόν ότι το Βιετνάμ δεν ε, βρίσκεται στον κατάλογο των χωρών που συστηματικά παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ούτε και στο, ε, ε, στην, στον κατάλογο των χωρών που χρήζουν ιδιαίτερης παρακολούθησης ή αρρωγής. επίσης, τα Ηνωμένα Έθνη ποτέ δεν έχουν εκδώσει από που να καταδικάζει ε, το Βιετνάμ. Επίσης, το Συμβούλιο ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, έχει εκδώσει 85 αποφάσεις για πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι για το Βιετνάμ. Καλούμε τις ευρωπαϊκές χώρες να συνεχίσουν να ε, να συνεχίσουν να ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τρίτο κύκλο αναθεώρησης ε, ε, του καταλόγου για, τα, το API για το 2019. Δεν έχετε άλλο χρόνο δυστυχώς. Δημερός με τα μέλη του Κοινοβουλίου μπορείτε να συνεχίσετε. Ο εισηγητής μας, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή που αφορά την ε, επικύρωση. Ε, οπωσδήποτε είχαμε εδώ μια πολύ σοβαρή ε, ανταλλαγή απόψεων, πρέπει να υπάρξουν και άλλες. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν σωστές αποφάσεις στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να επικυρωθεί η διαδικασία, γιατί πιστεύω ότι οι επιχειρήσει και από τις δύο πλευρές αυτό περιμένουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή τη στιγμή μια μοναδική ευκαιρία ε, να ειδωθεί ως global leader και ε, επανειλημμένα το είπαμε αυτό. Εδώ έχουμε μία μοναδική ευκαιρία ε, για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ίγκη και η ώρα. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή και δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν μια πρώτη συζήτηση στη διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσης πολλά και διάφορα συζητήσαμε. Οπωσδήποτε στο Κοινοβούλιο θα συνεχίσει η ε, μελέτη και η εξέταση των θεμάτων και των επιμέρους στοιχείων της συμφωνίας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι σήμερα ε, συνέλεξαν στοιχεία τα οποία θα πρέπει περαιτέρω να μελετήσουν. Ευχαριστώ πολύ σε όλους. Ευχαριστούμε τους εμπειρογνώμων.